So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die Plätze einzunehmen. Wir haben noch ein strammes Programm. Συνάδελφοι, καθίστε. Έχουμε μπροστά μας το πρόγραμμα για σήμερα το πρωί. Είχαμε τους ε, συντονιστές και είναι η τελευταία επίσημη συνεδρίαση της ομάδας στην τρέχουσα θετία. να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, αλλά στο 11 παρακαλώ να διευκρινίσω ότι θα ήθελα ε, να κοιτάξουμε ε, την έκθεση για την πρόληψη και διαχείριση των ξένων ειδών και στο σημείο 13 σε ό,τι αφορά την ε, τεχνική εφαρμογή των διατάξεων του Κιώτο, πολύ σημαντικές εκθέσεις που πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα την τελευταία στιγμή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τα κλείσουμε τα θέματα αυτά, αν συμφωνούν ε, οι συνάδελφοι να μπει στην ημερήσια διάταξη. Να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά τη διερμηνία έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από εστονικά και μαλτέζικα. Δεύτερη με ανακοίνωση έγιναν τριμερείς διάλογοι για τον έκθεση ε, για το Κιώτο 2 σε ό,τι αφορά τις τεχνικές εφαρμογές. Δευτέρα απόγευμα έγινε, υπήρξε συμφωνία με την Ελληνική Προεδρία και έτσι στο Παρίσι το 2015 στη διάσκεψη για το κλίμα αυτό θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των διαπραγματεύσεων. Στο σημείο 4 τώρα. Για τα πρακτικά λοιπόν έχουμε τις 30 Ιανουαρίου, τις 17 Φεβρουαρίου, 20 Φεβρουαρίου, 6 Μαρτίου και 10 Μαρτίου. Έχουμε όλα αυτά τα πρακτικά λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε σχόλια προσθήκες. Όχι. Ωραία, λοιπόν, θεωρούμε ότι εγκρίνονται ούτως τα πρακτικά. Και τώρα περνάμε λοιπόν στο σημείο 5 τέσσερα λέει ο πρόεδρος της ημερησίας διάταξη. Έχουμε ε, επισκέπτη από την Κοπενχάγη. Με μεγάλη μας χαρά τον υποδεχόμαστε. Χάν Μπράνιξ, εκτελεστικός διευθυντής ε, της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκού ε, Οργανισμού Περιβάλλοντος και θα ακούσουμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το πολιετές πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού. Εγώ το μόνο που μπορώ να συστήσω είναι να έχουμε στενές επαφές με την του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και αυτό και για τους νέους συναδέλφους γιατί έχουν μεγάλη τεχνογνωσία και πολλές γνώσεις για τις καθημερινές μας εργασίες. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο το είχα βάλει ως στόχο τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Ε, διατηρήσαμε στενές επαφές. Είναι ανεξάρτητοι οι οργανισμοί αυτοί. Δεν είναι εξαρτώμενοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματικά είναι κοσμήματα. Κοσμήματα αυτά που μπορούν να ε, ενισχύσουν την εργασία μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω ναι. άλλο, να δώσω με μεγάλη μου χαρά το λόγο στον Hans Μπράνεξ για να δούμε τι συμβαίνει μεταξύ του 2014 και του 2018 στη νέα εκτελεστική, στη νέα περίοδο. Uh, Ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση και για την πολύ ευγενική παρουσίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα σας παρουσιάσω το ε, πρόγραμμα εργασίας της επόμενης πενταετίας. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε δεν είχα ακόμη επιβεβαιωθεί στη θέση μου και χαίρομαι ακόμη περισσότερο που ξανασυναντιόμαστε σήμερα. Θα σας ε, παρουσιάσω λοιπόν το επόμενο πενταετές πρόγραμμα εργασίας που έχει εγκριθεί ήδη από το Διοικητικό μας Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις ε, προτάσεις των διαφόρων θεσμικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα εφαρμογή ε, του νέου προγράμματος εργασίας και θα έλεγα ότι από τα βασικά στοιχεία του σχεδίου εργασίας μας είναι ότι ε, προσπαθήσαμε να το ευθυγραμμίσουμε με τις κύριες πολιτικές των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι σημαντικό για τη συνοχή του έργου μας, αλλά λαμβάνουμε υπόψη και το μακροπρόθεσμο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κυρίως για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών. Βρίσκουμε την ισορροπία μεταξύ εφαρμογής των πολιτικών και μακροπρόθεσμων προοπτικών. Υποστηρίζοντας φυσικά τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας υπενθυμίσω ότι η αποστολή μας έχει μείνει και για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, την επόμενη πενταετία και παρέχουμε πληροφορίες σε οργανισμούς και φορείς λήψεων αποφάσεων και στο κοινό με ακριβή και αξιόπιστο τρόπο, στο μέτρο του δυνατού. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε σε σημαντικές και μετρήσιμες βελτιώσεις στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και ταυτόχρονα να, να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμά μας ε, το ευθυγραμμίζουμε με το πλαίσιο ανάπτυξη των πολιτικών γύρω από τα θέματα αυτά. Και φυσικά μας ενδιαφέρουν οι τομεακές πολιτικές του κοινοτικού κεκτημένου και θα συνεχίσουμε την παρακολούθηση και την ενημέρωση για την κατάσταση του περιβάλλοντος με πολλούς και διάφορους τρόπους στα πλαίσια των θεματικών πολιτικών. Επιπλέον λαμβάνουμε υπόψη την, ε, και πολύ σοβαρά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 με την προοπτική του 2030. Γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι περισσότερο περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών και θέλουμε να συμβάλλουμε στο θεματολόγιο αυτό υπό το πρίσμα των κλιματικών αλλαγών και του περιβάλλοντος. Επίσης είναι πολύ σημαντική η, η καινοτομία στη δημιουργία ε, λήψεων αποφάσεων ότι έχουμε την πολιτική αυτή σε, στα βασικά έγγραφα πολιτικής. Καταρχήν έχουμε το όραμά μας για μια κοινωνία με χαμηλή χρήση άνθρακα, μια προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων και ανθεκτικότητά τους και ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτά στα πλαίσια ε, μιας σταδιακής εφαρμογής των πολιτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Θέλουμε να γίνουμε η πρωταρχική πηγή γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές. Θεωρούμε λοιπόν ότι η εφαρμογή είναι πολύ σημαντικό θέμα και βρίσκεται στο επίκεντρο των στόχων μας. Θέλουμε να γίνουμε ε, ένα ε, κέντρο γνώσης και Αναφέρεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ότι υπάρχει κενό της γνώσης και χρειάζεται ενίσχυση των γνώσεών μας. Εμείς λοιπόν επικεντρωνόμαστε στο, στην πτυχή γνώση στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Θέλουμε να πρωτοστατήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να διευκολύνουμε την ανταλλαγή των γνώσεων και τη δημιουργία ικανοτήτων, κάτι που σε μεγάλο βαθμό θα χρησιμοποιήσει το, το δίκτυο που έχουμε δημιουργήσει με τα κράτη-μέλη και που είναι ε, απαραίτητο για τη λειτουργία μας. Το AONET που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον. Τώρα θέλουμε να, να συνδέσουμε το θέμα περιβάλλον και κλιματικές αλλαγές με τις α, ε, βασικές πρωτοβουλίες μας και το SOER, την... Ε, αξιολόγηση, την εκτίμηση βιωσιμότητας και τις εκθέσεις κατάστασης για το περιβάλλον. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι το 2015 θα ολοκληρώσουμε το ΣΟΕΡ αυτή την εκτίμηση βιωσιμότητας και αναφορά στις κατάσταση του περιβάλλοντος προκειμένου ε, να μπορέσουμε να σας δώσουμε πριν το τέλος του 2014 και με, την, ε, με το νέο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουμε να σας τροφοδοτήσουμε με πληροφορίες ώστε το 2015 να έχουμε ανταλλαγές απόψεων με τις χώρες μέλη, με εσάς και με άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα για τα πορίσματα που έχουμε συγκεντρώσει και τις γνώσεις που έχουμε συγκεντρώσει την τελευταία πενταετία. Το ΣΟΕΡ του 2015, εκτίμηση δηλαδή βιωσιμότητας και ενημέρωση κατάστασης του περιβάλλοντος, θα λάβει υπόψη και, την, και το μεταβατικό θεματολόγιο. Τώρα, ο τίτλος του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον είναι το FZIN, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τα οικολογικά όρια. Τα λαμβάνουμε υπόψη πολύ σοβαρά, τα οικολογικά σύνορα, τα οικολογικά όρια, που θα μας περιορίσουν στον 21ο αιώνα. Βλέπουμε τα διάφορα οικολογικά συστήματα, το ενεργειακό σύστημα, το επιστηστικό σύστημα, το, το σύστημα κινητικότητας, όλα αυτά τα συστήματα θα, θα χαρακτηρίσουν ε, τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές. Έχουμε την, ε, το θεματολόγιο για την πράσινη ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη. Όλα αυτά θα πρέπει να λάβουν χώρα στα όρια των οικοσυστημάτων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ενοιολογικά όρια που θα επεξεργαστούμε στην επόμενη πενταετία. Φυσικά ε, είχαμε μέχρι τώρα δύο δεκαετίες επενδύσεων. Μέχρι το Μάρτιο του 2015 μας ε, αξιολογούσε ανεξάρτητα η COE και αποτέλεσμα είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι ε, πιο αποτελεσματική και αποδοτική λύση για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για την κατάσταση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντο. Είχαμε μέχρι στιγμή δηλαδή πολύ θετικέ αξιολογήσει από αυτόν τον ανεξάρτητο φορέα το COWI. Έχουμε εντοπίσει τέσσερι ε, τομεί στρατηγική ε, για το πρόγραμμά μα. Θα του αναλύσω εντό ολίγου. Και μάλιστα θέλουμε να υιοθετήσουμε αυτού του τομεί στρατηγική για να συμβάλλουμε στον γενικό κύκλο των πολιτικών. Δεν καταμετρούμε απλώς, δεν αξιολογούμε, δεν παρακολουθούμε και δεν υποβάλλουμε εκθέσεις για το περιβάλλον κατόπιν ορτής, δηλαδή μετά την εφαρμογή των πολιτικών, αλλά θέλουμε στο μέλλον να εντοπίζουμε και νέα θέματα, να κάνουμε μια πλαισίωση των θεμάτων στο επόμενο πρόγραμμα δράσης και επίσης να εντοπίζουμε μέτρα πολιτικών και ανάπτυξη πολιτικών ώστε να συμβάλλουμε με τις γνώσεις μας στη διαμόρφωση των πολιτικών. Τώρα, ο, πρώτο ο πρώτος στρατηγικός τομέας είναι η ενημέρωση για την εφαρμογή της πολιτικής. Θέλουμε να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, την προσπελασιμότητα και τη χρήση ε, των ε, πληροφοριών για το περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσθέτουμε πληροφορίες στο ευρύτερο πακέτο πεδίο εφαρμογή δηλαδή, αλλά και θέλουμε όλο και μεγαλύτερη και καλύτερη ποιότητα και συμπερίληψη πιο συστημικών πληροφοριών και βελτίωση της πρόσβασης σε όλες τις διαπαφές τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών. Και αυτό το κάνουμε σε... με βάση τα πάγια πλαίσια που έχουμε, αλλά και υπό το φως των νέων θεμάτων. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την ενημέρωση και την υποβολή εκθέσεων, όπως κάνουμε και στο παρελθόν, με ποιοτικέ εκθέσεις. Τα νέα θέματα που θα είναι προτεραιότητες στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού ε, συνάδουν με τις προτεραιότητες του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Καταρχήν, ε, ατμοσφαιρική ρήπανση, μεταφορές και η Δεύτερο τομέα είναι η βιομηχανική ρήπανση και μάλιστα δημιουργήσαμε και ένα, μια νέα ομάδα εργασία. Θέματα περιορισμού των κλιματικών αλλαγών και ενέργεια, αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών τροτότητα και προσαρμογή, διαχείριση του ύδατος πόρων και οικοσυστημάτων, θαλάσσια και ναυτιλιακή πολιτική αλία και παράκτιες περιοχέ, βιοπικιλότητα, οικοσυστήματα, γεωργία και δάση, ε, αστικός, ε, αστικό περιβάλλον, χρήση γης και εδάφους και τέλος ε, απόβλητα και πόροι από υλικά. Και μάλιστα οι, πόροι από τα υλικά αυτά ίσως θα είναι και το μέλλον, το επίκεντρο στην μελλοντική ατζέντα μας πολύ περισσότερο από την διαχείριση ή την ε, επεξεργασία αποβλήτων. Τώρα, θέλουμε να συμβάλλουμε στη, στην υποβολή εκθέσεων ε, με βάση την επιτροπολογία και τις πολυμερείς συμφωνίες και να υποβάλουμε εγκαίρως ε, με βάση δεδομένων, δείκτες και άλλες μορφές επικοινωνίας. Δεύτερος στρατηγικός τομέας προβλέπει την εκτίμηση των συστημικών προκλήσεων. Τα τελευταία 10 με 15 χρόνια ασχολούμαστε με τη βελτίωση ολοκληρωμένων αξιολογήσεων προκειμένου να εντοπίσουμε συνέργειες και να στηρίξουμε τη συνοχή των πολιτικών. Και μάλιστα αυτός ο στόχος, αυτός ο τομέας εντάσσεται και στην ατζέντα των πολιτικών, ώστε να έχουμε πιο συνεκτικές πολιτικές. Θα κάνουμε και αναλύσεις προβλέψεων προκειμένου να εντοπίζουμε νέα θέματα. Το κάναμε και στο παρελθόν, θα το συνεχίσουμε σε συστημικό επίπεδο και θέλουμε να παρέχουμε γνώση και ανάλυση για να εκτιμηθεί η πρόοδος προς ε, θεμελιώδεις ε, μεταβάσεις. Και μάλιστα μια γραφική παράσταση που χρησιμοποιείται συχνά όταν μιλούμε για μετάβαση είναι ότι όταν έχουμε σωστές πολιτικές μακροπρόθεσμα θα περάσουμε από μια κατάσταση μη βιώσιμη προς όλο και βιωσιμότερη κατάσταση. Αυτή είναι βέβαια μια πολύ αισιόδοξη θεώρηση της κατάστασης. Άλλη δυνατότητα είναι να εξασφαλίσουμε σοβαρή ανάλυση και συγκέντρωση γνώσης. Γιατί θα μπορούσαμε να προσκρούσουμε σε αδιέξοδα. θα μπορούσαμε να δαπανούμε πολλά κονδύλια στην Ευρώπη και να εγκλωβιζόμαστε όλο και περισσότερο τα παρόντα συστήματα για την κινητικότητα, για την ενέργεια, για τα τρόφιμα και μάλιστα το 2020, ακόμη και το 2030 να είμαστε ικανοποιημένοι με την υλοποίηση των στόχων, αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε ε, είτε μένοντας εγκλωβισμένοι στα τρέχοντα συστήματα, είτε υιοθετώντας μια πιο ανοιχτή στάση προς μελλοντικά συστήματα. Φυσικά εμείς χρησιμοποιούμε τη γνώση ως βάση και θέλουμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι ένα ε, αποτέλεσμα boomerang, Δηλαδή να μην εθετήσουμε πολιτικές ε, σήμερα που μετά από μερικά χρόνια θα μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ήταν ακατάλληλες και ότι δεν ε, μας επέτρεψαν να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και ότι γυρίζουν σαν boomerang. Φυσικά θέλουμε ένα σύστημα που θα στηρίζεται στη γνώση και να αποφύγουμε οποιαδήποτε κατάρρευση του. Τώρα, εκτίμηση των συστημικών προκλήσεων. Αυτό θα το κάνουμε ε, αναλύοντας την οικονομία που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και το περιβάλλον. Μας ενδιαφέρει η πράσινη ατζέντα και η πράσινη ανάπτυξη. Επίσης, σε συνδυασμό με τη Eurostat, τον ΟΣΑ και άλλους φορείς εξετάζουμε αυτό το θεματολόγιο. Μας ενδιαφέρει φυσικά το περιβάλλον, η ανθρώπινη υγεία και ευημερία για παράδειγμα χημικές ουσίες και ανθρώπινη υγεία και ο συσχετισμός τους. Ε, συνεργαζόμαστε με το JRC για θέματα υγείας και περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πολιτικές της ε, κινείται σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οπότε οι μέγα τάσεις μας ενδιαφέρουν για να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για μετάβαση και Αυτά όλα στα πλαίσια του, της εκτίμησης βιωσιμότητας και έκθεσης κατάστασης του περιβάλλοντος για το 2015 εν ώψη του 2020. Και θα πρέπει να κάνουμε και μια τακτική αξιολόγηση του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, οπότε θα δίνουμε συνεχώς τα αποτελέσματα στα επόμενα χρόνια και στο επόμενο περίοδο, δηλαδή 2014 με 2018. Γίνεται εβδομαδία αξιολόγηση της ε, φάσης στην οποία βρισκόμαστε για το ΣΟΕΡ σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Παρέχουμε εκθέσεις, ε, ετήσιες εκθέσεις για τους δείκτες και έχουμε και την ε, online πλατφόρμα SOE, δηλαδή συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση των πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη με συμπερίληψη των πιο πρόσφατων στοιχείων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιοι φορείς αλλά και το κοινό. Και φυσικά συνεχής αξιολόγηση του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Τώρα θέλουμε να συμβάλλουμε στην παραγωγή γνώσης, ανταλλαγής και χρήσης. Θέλουμε να γίνουμε αυθεντία και κόμβος γνώσης και πληροφοριών στην Ευρώπη και να συμβάλλουμε στην ε, δημιουργία γνώσης και στην κατανομή της, στην ανταλλαγή της και τη χρήση της. Έχουμε μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη και τεράστιο δίκτυο. Είμαστε ασυναγώνιστοι στον κόσμο και έχουμε πολύ στέρεη βάση εργασίας. Βέβαια ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε σεμνοί λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μα και δεν θέλουμε να είμαστε απομονωμένοι, αλλά να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς και παράγοντε. Τώρα πώς ε, το επιδιώκουμε. Χρησιμοποιούμε το δίκτυο AONET, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρηση και Παρατήρησης για το Περιβάλλον. Έχουμε βέβαια και εταιρικέ σχέσει με Βορρά και Νότο και δίκτυα γραμματείες ε, επιμέρους οργανισμών περιβάλλοντος. Έχουμε ανεπτυγμένο δίκτυο και χρησιμοποιούμε τα τεχνικά συστήματά μας, την ανταλλαγή γνώσεων και την παραγωγή γνώσης. Επίσης έχουμε αγαστή συνεργασία με τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Έχω ε, πολύ σημαντική επικοινωνία στο εγχείρημα αυτό. Βέβαια, η επικοινωνία δεν περιορίζεται στις δημόσιες σχέσεις, αλλά στην στενή συνεργασία με τους εταίρους μας. Ποιοτική διαχείριση επίσης είναι πολύ σημαντικό και διαχείριση πληροφορίας ε, επίσης σημαντικός τομέας. Αυτή τη στιγμή μάλιστα έχω μία νέα συμφωνία ε, με την DGR, τη, τη, τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και τις ε, υπηρεσίες του Κοπέρνικος ώστε να παρέχουμε και σε αυτές ε, περιβαλλοντικές υπηρεσίες ε, για τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά συνδέονται με, την με τις βασικές διαδικασίες ε, του ΕΟΠ με το ΕΙΟΝΕΤ. Δηλαδή, συγκεντρώνουμε δεδομένα και στοιχεία από μια πληθώρα πηγών. Έχουμε και μια διασύνδεση με τη διαδικασία του ορίζοντας 2020 και τις ερευνητικές προσπάθειες. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το RTD για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις μαζικές επενδύσεις που γίνονται σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Έτσι έχουμε πολύ καλύτερα δεδομένα και δημιουργούμε καλύτερους δείκτες και βάσεις δεδομένων κάνουμε καλύτερες αξιολογήσεις, πιο εμπεριστατωμένες και ενισχύουμε τη βάση γνώση που, χρειαζόμαστε και για το 7ο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον, αλλά και για τα μακροπρόθεσμα προγράμματα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη συμπαραγωγή γνώσης, ανταλλαγή και χρήση της, τι θέλουμε, να ενισχύσουμε το AONET, θέλουμε μετρήσεις για την καταμέτρηση της ενεργού συμμετοχής του Aionet ε, online παροχή των δεδομένων του ΕΟΠ σε υψηλό επίπεδο και επίσης ε, κάνουμε προσπάθειες ε, επικοινωνίας και θέλουμε να δούμε τι αποτελέσματα έχουν. Βέβαια, η διαχείριση του ΕΟΠ ε, είναι στρατηγική σημασία και εκεί ο στόχος μας είναι απλούστατος. Αριστεία στην εκτέλεση του προγράμματος εργασίας μας. Δηλαδή δίνουμε έμφαση ιδιαίτερη στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση και εννοείται και στην διοίκηση και τη συμμόρφωση με όλους τους κανόνες που ισχύουν και για το δικό μας οργανισμό. Θέλουμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα εργασιών και να έχουμε θετικό αποτέλεσμα στην επόμενη αξιολόγηση των εργασιών μας. Εν κατακλείδη, Θεωρώ ότι η φιλοδοξία μας είναι να συνδέσουμε στο έργο μας τους τρεις χρονικούς ορίζοντες ε, που σας ανέφερα στην αρχή, δηλαδή να συνεχίσουμε την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του κοινοτικού κεκτημένου σε καθημερινή βάση, αλλά να το συνδέσουμε και με την ε, στρατηγική και το πρόγραμμα για το 2020, το 2030 και το θεματολόγιο για το 2050, κάτι που προϋποθέτει καινοτομία στην δημιουργία γνώσης. Έχουμε λοιπόν διάφορες εσωτερικές διαδικασίες και συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς. Βέβαια η Ευρώπη αυτό το, κα... έχει... το κάνει και επιτελεί το έργο του σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο. Έχουμε επίγνωση ότι ξεκινούμε μια πενταετία περικοπών στον προϋπολογισμό και λιτότητας, οπότε σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να επανειεραρχήσουμε τους πρωταρχικούς μας στόχους και αυτό θα γίνει στο πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας. Και έχουμε εδώ δύο προσεγγίσεις ε, για τις περικοπές ε, στο προσωπικό και τον προϋπολογισμό. Η μία προσέγγιση είναι να καθίσουμε σε μια γωνίτσα και να κλαίμε τη μοίρα μας και να κατηγορούμε τους αρμόδιους για τον προϋπολογισμό, αλλά δεν είναι αυτή η μυρολατρεία ή το πάθεια χαρακτηριστικό μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε διορατικοί, αισιόδοξοι και θετικοί. Νομίζω ότι έτσι θα κρατήσουμε αμύωτο τον ενθουσιασμό μας και ως οργανισμός, αλλά θα επιτρέψουμε και την ε, σωστή πορεία προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτά σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για να λύσω απορίες σας. Σας ευχαριστώ πάντως για την ευκαιρία που μου δώσετε να σας παρουσιάσω το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπράνεγκς για, τις, ε, για την παρουσίαση αυτή και έχω κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα ωστόσο να δώσω το λόγο πρώτα στο άτομο επαφής μας και να σας ευχαριστήσω που ε, είναι εδώ ε, έχουμε τον κύριο Γκερμπράντι εδώ και πάντα διατηρεί λοιπόν τις επαφές με, την, ε, με τον οργανισμό. Ο κύριος Γκερμπράντι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ήμουν ε, πραγματικά, ήταν τιμή μου και προνόμιό μου που ήμουν το άτομο επαφή με τον οργανισμό, γιατί αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ πιο στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο, να αξιοποιήσω τι γνώσει αυτέ πιο πολύ. Κάποια σχόλια και κάποιες παρατηρήσεις, επιτρέψτε μου. Καταρχάς, κύριε Μπράνεξ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση του πολυετούς προγράμματος εργασίας. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό σας. Αναφερθήκατε στα τελικά σας συμπεράσματα ότι υπάρχουν περιορισμοί ασφαλώς ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι εν γέννη για οποιαδήποτε οργανισμό είναι καλό να χρειάζεται να εξετάζει εντελεχώς ε, τον προπολογισμό του. Έχετε όμως πουθενά την αίσθηση ότι τα επόμενα χρόνια σε κάποιους τομείς δεν θα έχετε επαρκή χρηματοδότηση για να εκτελέσετε τα καθήκοντα τα οποία σας έχουμε αναθέσει ως νομοθέτες. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μου ερώτηση. Έχετε λοιπόν την αίσθηση ότι ο προϋπολογισμός για τα επόμενα έτη επαρκεί για το τεράστιο όγκο καθηκόντων που έχετε. Δεύτερη παρατηρήση, ερώτηση, αν θέλετε, και πρόταση, σύσταση προς την Επιτροπή μας. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο την γνώση που έχει ο οργανισμός σας και το όλο δίκτυο το οποίο συνοδεύει. Μιλάμε για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και πολύ συχνά αναφέρουμε ότι Υπάρχει μεγάλος όγκος γνώσης που αναπτύσσεται. Ωστόσο, συχνά το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν, δεν αντιλαμβάνονται ενδεχομένω και πάντα τον τεράστιο όγκο γνώσης που υπάρχει. Και έχω την αίσθηση ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και εδώ, και εδώ δηλαδή στο Κοινοβούλιο ως εισηγητής έχω διοργανώσει και για την βιοτυπικιλότητα και για την ενεργειακή αποδοτικότητα μια ολόκληρη ημερίδα εδώ στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους του οργανισμού για να συζητηθούν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές όλων αυτών των θεμάτων. Αμφιβάλλω όμως αν το κάνουν αυτό και άλλοι συνάδελφοι. Ρωτώ λοιπόν και εσάς αλλά και τη γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τη γνώση του οργανισμού σας στην Κοπενχάγη. Θεωρώ ότι μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα λοιπόν αυτή η πηγή γνώση. Ίσως λοιπόν θα πρέπει από κοινού να αναζητήσουμε τρόπους καλύτερης αξιοποίησης της γνώσης αυτής. Ε. Αυτό το απευθύνει και ω ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, διατηρείται εξαιρετικές σχέσεις με την Γενική Διεύθυνση, Κλίμα, Ένβη και το καθεξής. Διαβάζοντας όμως το άρθρο σας στο website του ΕΟΠ για τις συστημικές προκλήσεις και ότι δεν θα πρέπει να πρασινίσουμε, να δώσουμε πράσινο χαρακτήρα σε κάποιους μόνο τομείς της οικονομίας, αλλά σε όλη την οικονομία, αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτό να το προωθήσουμε ως μήνυμα προς τη Γενική Διεύθυνση Enterprise Επιχειρήσεων, γιατί μπορούμε να επιμένουμε στα θέματα αυτά ε, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβούλου, στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή, αλλά τελικά η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων τελικά καθορίζει την πορεία της οικονομίας. Καλύτερα λοιπόν αξιοποίηση των γνώσεων του οργανισμού σας χρειαζόμαστε. Κατά τρίτον, επικεντρώνεστε σε θέματα εφαρμογής. Πολύ σωστά αποτέλεσε άλλωστε και τον πυρήνα των προτεραιοτήτων του Επιτρόπου Ποτόσνικ πριν από κάποια χρόνια που ξεκίνησε. Τεράστιο πρόβλημα αυτό ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη υστερούν σε θέματα ε, μεταφορά τη νομοθεσία και έχω την αίσθηση ότι του απασχολεί όλο και λιγότερο το θέμα αυτό σε σχέση πριν από, πριν από κάποια χρόνια. Το πρόβλημα οξύνεται. Δεν αμβλύνεται. συζητήσαμε ενδεχόμενε ευρωπαϊκέ επιθεωρήσεις για θέματα εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή νομοθεσίας και σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό θέμα. Πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό και ιδιαίτερο τώρα, ξέρετε, με τα αντιευρωπαϊκά συναισθήματα και τι αντιευρωπαϊκέ δυνάμει που αναδύονται όλο και πιο πολύ. Ο οργανισμός σας, έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρω ότι διστάζει να θέσει το θέμα των επιθεωρήσεων. Αλλά πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερο ρόλο να αντιδραματίσει ο οργανισμός σας. Τέλος, τελευταίο ερώτημα για την ε, αποδοτικότητα των πόρων. Με χαροποιεί αυτό που αναφέρετε στο πρόγραμμα εργασία σας για την ε, αποδοτικότητα των πόρων. Έχετε πολύ σωστούς στόχους για την αποδοτικότητα, για τους στόχους. Για το χρονοδιάγραμμα όμως, τι γίνεται νέες μελέτες προετοιμάζονται για τα επόμενα χρόνια, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα για την ενεργειακή επιδοτικότητα της οποίας προεδρεύει ο Επιτροπός Ποτόσνικ, ε, αναπτύσσονται τέτοιοι στόχοι. Υπάρχει δυνατότητα να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία προκειμένου να είμαστε και πιο συντονισμένοι με τις Βρυξέλλες προκειμένου να μην ε, δημοσιεύσετε τις συστάσεις σας αφότου έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ τον κύριο Γερμπράντη να πω ότι συμφωνήσαμε με τον Γενικό Διευθυντή του οργανισμού να διοργανωθεί ένα σεμινάριο στην αρχή της επόμενης θητείας και για τους βοηθούς των νέων ή των παλιών συναδέλφων και για, τα ίδια, τους ίδιους τους βουλευτές για να ξέρουμε ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία της εργασίας του οργανισμού. Θέλω να τονίσω ότι είναι τεράστιο όγκο των ε, γνώσεων που έχουν συσσωρευτεί και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο θέμα των, της συνεργειακής αποδοτικότητας. Συμφωνήσαμε στους συντονιστές να προωθήσουμε το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αποδοτικότητας των πόρων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έχουμε συγκεκριμένες προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πολλά είχαν ε, ανακοινωθεί και εδώ και ένα, ένα μισή έτος έχουμε τελματώσει πλήρως αυτό λοιπόν είναι παράδεκτο. Επόμενος ομιλητής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λούντον ο οποίος είναι εδώ σήμερα να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία για να του δώσουμε το λόγο. Και ο κύριος Χολσπέικ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως ένας από τους εκπροσώπους αυτής της Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν έχω πολλές παρατηρήσεις να κάνω. Ο Οργανισμός της Κοπενχάγης παρασμένει στη ε, ε, ανώτερο, στην ανώτερη ιεραρχία όσον αφορά την απόδοση. Η έρευνα την οποία ε, προβαίνει είναι υψηλότατου επίπεδου. Ε, έχουμε εξαιρετικές δυνατότητες και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το τι κάνει αυτός ο οργανισμός. Έχω δύο μικρές παρατηρήσεις να κάνω. Δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών και της περιορισμού ορισμένων θεμάτων πρέπει να προβούμε σε κάποιες επιλογές και λυπούμε διότι φαίνεται ότι η εργασία της Επιστημονικής Επιτροπής φαίνεται να υποβαθμίζεται Πιστεύω πως είναι σημαντικό όχι μόνο για τον οργανισμό αλλά και για το Ευρωκοινοβούλιο η Επιστημονική Επιτροπή η οποία είναι ένας πολύ, ένα πολύ καλό σύνολο Ευρωπαίων επιστημόνων να μπορεί να κάνει την δουλειά της όπως ε, πρέπει διότι εάν πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο βαθμό δραστηριότητας χάνεις το νόημα της ύπαρξής σου. Επίσης το να εντοπίζουν ε, αναδυόμενα θέματα να εξασφαλίζουν τις προτεραιότητες και την απόδοση των προγραμμάτων όπου η Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να παίξει πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο χωρίς Επιστημονική Επιτροπή το να γίνει μια συζήτηση ας πούμε για τα βιοκαύσιμα με το, μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα είχε ποτέ την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα των βιοκαυσίμων τόσο εις βάθος και τόσο έγκαιρα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η Επιστημονική Επιτροπή να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται όπως πρέπει. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ευαίσθητο θέμα όπου νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς το IONET θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης και Παρατήρησης σχετικά με το περιβάλλον δεν ε, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη σχετική δραστηριότητα. Αυτό, γι' αυτό με λυπεί. Πρέπει να σκεφτούμε αν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους εκεί και ίσως Μάλιστα και να πρέπει να διοργανωθεί το AONET εδώ στις Βρυξέλλες ώστε και ε, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούν να πάνε ως παρατηρητές και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι πιο κοντά. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Χόλσπεκ. Να το είναι τώρα να δώσουμε το λόγο στους συντονιστέ ε, όπως ήθιστε, και να απαντήσει στη συνέχεια ο κύριο Μπράουνινγκς και μετά να πάρουν το λόγο και οι υπόλοιποι ε, ε, συνάδελφοι. Ο Ρίχαρτ Σέμπερ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά και τις δραστηριότητε της. Δύο ε, ερωτήσεις, μία πιο συγκεκριμένη. Τι κάνει συγκεκριμένα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος για να υπάρχει πιο ενιαία διαχείριση των δεδομένων. Ξέρετε ότι όταν αλλάζουν κάποιοι κάποιες τρόπο συλλογή των ε, στοιχείων μπορεί να αλλάξει και το αποτέλεσμα. Αυτό έχει να κάνει και με την οικονομία. Θα πρέπει να είναι όμως ενιαία τα στοιχεία, γιατί στην περίπτωση αυτή είναι πιο ε, σαφή και πιστικά τα αποτελέσματα που προβάλλονται. Πώ λοιπόν... Ε, ξέρετε, αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, η οικονομία γενικά. Πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε ένα ενιαίο χαρακτήρα σε αυτά τα στοιχεία τα δεδομένα προκειμένου να είναι και κοινή η αξιολόγηση, η εκτίμησή τους, η χρήση τους. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις ε, αντιμετωπίζουμε πολλές διαφορετικές εμπειρογνωμοσύνες και ε, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που καταλήγουν σε αντιδημητρικώς ε, αντίθετα αποτελέσματα. Δεύτερη ερώτηση. με ποια μοντέλα μπορείτε να προσαρμόζεστε στην ταχαίως μεταβαλλόμενη τεχνολογική εξέλιξη. Πώς μπορείτε λοιπόν αυτή την τεχνική μεταβολή, αυτή την τεχνική αλλαγή που είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις στις προβολές σας, πώς ε, την λαμβάνετε υπόψη, πώς την ε, εντάσσετε στις προβολές σας σε ό,τι αφορά την έρευνα, τις εξελίξεις, αλλά και την τεχνική συγκεκριμένη εφαρμογή. Και μία συγκεκριμένη ερώτηση. Ήμουν εισηγητής σε ό,τι αφορά τις ε, ουσίες προτεραιότητας και όπως ξέρετε ε, τέθηκαν ε, το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα φαρμακολογικά προϊόντα στο νερό, σε ό,τι αφορά την συλλογή δεδομένων και σε ό,τι αφορά την φαρμακευτική στρατηγική. Πώ μπορούμε λοιπόν να την εντάξουμε αυτή τη στρατηγική σε ό,τι αφορά και αυτά τα δεδομένα αυτή, γιατί θεωρώ ότι αυτό επηρεάζει και την πολιτική των φαρμακολογικών εταιριών, αλλά και την ίδια την πολιτική. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πρόεδρος. Chris σύντομα. Νομίζω ότι στις παρατηρήσεις σας καταστήσατε αρκετά σαφές πως ο οργανισμός επιθυμεί να αναμειχθεί στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Κομισιόν. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι η Κομισιόν εισακούει τις προτάσεις της, του οργανισμού όσο θα έπρεπε για συγκεκριμένα μεμονωμένα θέματα. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη σχέση και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως ο ε, οργανισμός έχει τον κατάλληλο την κατάλληλη επιρροή δεδομένων των πόρων που του χορηγούμε. Και δεύτερον, Εάν δούμε τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε η Κομισιόν τα τελευταία πέντε χρόνια, εγώ τώρα εδώ έχω υπηρετήσει τρεις θητείες και θυμάμαι, ε, θυμάμαι να ε, μας πλημμυρίζουν οι νομοθεσίες κάθε θητεία. Τα τελευταία όμως θητεία, παρά το γεγονός ότι έχουμε δουλέψει σκληρά, όπως λέει και ο Πρόεδρος, ε, είχαμε αρκετή ησυχία ας πούμε νερό, αέρας, ναι, ήταν θέμα αναθεώρησης, αναδιατύπωσης. Σε τι οφείλεται αυτό, θεωρείτε ότι λείπει ακόμα πρωτογενής νομοθεσία ή θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στις δράσεις επιβολής και εξασφάλισης της σωστής εφαρμογής αυτών των νομοθεσιών ή στις ε, εθελοντικές συμφωνίες που δυστυχώς στο παρελθόν δεν ήταν αποτελεσματικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώσαμε τους ε, συντονιστές και έτσι λοιπόν θα ήθελα να κλείσω τον πρώτο γύρο ερωτήσεων, να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Μπράνιξ να απαντήσει. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας και για τις συστάσεις σας ε, ακόμη. Θα τις ανατρέξω καταρχήν για να απαντήσω στον κύριο Γερμπράντη για τον προϋπολογισμό. Έχουμε κάνει τις προβλέψεις μας για το τι μπορούμε να κάνουμε με βάση μια υπόθεση ισόπεδου προπολογισμού, λόγω του πληθωρισμού δηλαδή, ο προπολογισμός μας θα μειωθεί γύρω στο 10% στην ουσία. Έπειτα πρέπει να λάβουμε υπόψη περιορισμούς στο ανθρώπινο δυναμικό, όπου το οργανόγραμμά μας θα καθοριστεί ανάλογα με το τι θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες. Ο συνδυασμός ε, αυτών των δύο μάλλον θα σημάνει ουσιαστικές περικοπές στο προσωπικό μας. Αυτό επηρεάζει το τι κάνουμε, αλλά και το πώς το κάνουμε. Τώρα, πώς το αντιμετωπίζουμε. με δύο τρόπους. Αν και δεν έχουμε γράψει στο έγγραφο ρητά το τι υποβαθμίζεται και τι όχι, υπάρχουν πολύ ρητές επιλογές στο έγγραφο που περιγράφονται όντως θα χάσουν την έμφαση τους κάποια θέματα, την ε, προτεραιότητά τους και θα μείνουμε πιο κοντά στις κεντρικές μας δραστηριότητες. Επίσης θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε με ευφιέστερο τρόπο, εμπλεκόμενοι στα δίκτυα με διαφορετικό τρόπο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε παίξει δραστήριο ρόλο στο πανευρωπαϊκό πανόραμα μέσω των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Ευρώπη. Έχουμε επίσης εμπλακεί σε διάφορες παγκόσμιες διαδικασίες και θα προσπαθήσουμε αυτό να το κάνουμε με πιο αποτελεσματικό για τους πόρους μας τρόπο. Δηλαδή δεσμευόμενοι σε ευρωπαϊκές συμβολές υψηλής ποιότητας για όλα αυτά τα θέματα, γιατί αυτός είναι ο βασικός μας κεντρικός μας ρόλος, αλλά και καλώντας άλλους να μάθουν από τη δική μας εμπειρία και όχι να είμαστε υπομπή αυτής της εμπειρίας η αγγελιοφόροι ε, και να φτιάχνουμε δυνατότητες αλλού στον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εστιάσουμε σε ποιοτικέ συμβολές και στις ουσιαστικές πτυχές της διαδικασίας. Επίσης ε, θα ε, μειώσουμε σημαντικά τα επόμενα χρόνια τον προπολογισμό μας όσον αφορά τις αποστολές. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να φτιάχνουμε συναντήσεις που να μην απαιτούν ταξίδια μετακινήσεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνουμε εξοικονομήσεις, αλλά τελικά νομίζω πως ναι, θα χρειαστεί να κάνουμε και επιλογές. Έχουμε δεσμευθεί στο να το παρακολουθούμε όλα αυτά με διαδραστικό τρόπο εσωτερικά. Είναι στην ημερήσια μας διάταξη. Η διευθυντική μας ομάδα ασχολείται διαρκώς με το θέμα και για οποιαδήποτε μας επιλογή για αντικατάσταση κάποιου ή για αντικατάσταση ή για μετάθεση ή για αποχώρηση θα, θα πολύ σοβαρά υπόψη τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους είναι ο βασικός μας, η βασική μας, ε, με το βασικό μας μέλημα. Δεν είναι βέβαια το πιο ευχάριστο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε στο προσωπικό μας. Είναι επίσης κάτι το εντελώς νέο, γιατί ο οργανισμός τα τελευταία 20 χρόνια μόνο αυξήσει προσωπικού είχε δει και αυξήσεις προϋπολογισμού. Θα πρέπει επίσης να δούμε ότι ε, επιπλέον έχουμε παραπάνω δουλειά. Επίσης ο κ. Κερμπράντη ρώτησε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα νέα μας καθήκοντα τα επόμενα χρόνια. Πώς ξέρετε, Έχω η Ευρώπη έναν μηχανισμό για τα νέα καθήκοντα και υπάρχει ένας μηχανισμός για την πρόσληψη προσωπικού που συνδέεται με τα νέα καθήκοντα. Θα χρειαστεί να, ε, λοιπόν να συνεργαστούμε με την Κομισιόν ώστε να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους όταν έχουμε νέα καθήκοντα. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν μπορούν να προσθεθούν πολλά επιπλέον καθήκοντα χωρίς νέους πόρους, γιατί πραγματικά είμαστε πολύ στριμωγμένοι. Καλύτερη γνώση και επικοινωνία. Ορισμένοι ρώτησαν για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν τρόποι να βελτιωθούν όλα αυτά. Καταρχήν ο χρονισμός. Τα τελευταία χρόνια ένα πολύ καλό παράδειγμα για τον συγχρονισμό της επικοινωνίας που βοήθησε τη διαδικασία της συγκρότησης πολιτικής ήταν οι αναθεωρήσεις μας, τα review μας ε, πραγματικά προσπαθήσαμε να συντονιστούμε τις Βρυξέλλες για το πότε πρέπει να δίνουμε τις πληροφορίες μας αλλά και με ποια μορφή γιατί έχουμε μια ολόκληρη σειρά από εκθέσεις αλλά δεν είναι πάντοτε και ευκο, ευανάγνωστες για τους ηθήνοντες της πολιτικής και γι' αυτό και ε, εργαζόμαστε για διάφορες μορφές αποστολής μηνυμάτων, όπως ας πούμε γραφήματα, ε, πλαισίωση των θεμάτων. Ε, να μην έχουμε δηλαδή σελίδες επί σελίδων που πιάνουν ολόκληρα τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά πιο άμεσα μηνύματα. Τι σημαίνει αυτό ας πούμε για τα κοινωνικά συστήματα, τι σημαίνει αυτό για τη σύνδεση των πολιτικών με τις οικονομικές πολιτικές, τι σημαίνει για την υγεία. Προσπαθούμε δηλαδή να συντάσσουμε έτσι τα μηνύματά μας ώστε να είναι πιο εύληπτα ε, για τους ε, πολιτικούς ε, ηθήνοντες. Επίσης, προσπαθούμε να τροποποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σας στέλνουμε εσάς πληροφορίες. Παλιότερα ήταν πιο σκόρπια τα πράγματα, σας ενημερώναμε για οτιδήποτε κάναμε. Ενώ τώρα είμαστε συνδεδεμένοι μέσω ενός πιο προηγμένου συστήματος, όπου μπορείτε να μας υποδείξετε τι είδους πληροφορίες θα θέλατε να παίρνατε. Επίσης, ε, στη συνέχεια έχουμε τις επισκέψεις ε, που ε, γίνονται στον οργανισμό, που είχαμε το περασμένο φθινόπωρο επίσκεψη του Κοινοβουλίου. Θα σας καλέσουμε φυσικά και πάλι και ελπίζουμε να σας δούμε στην Κοπεχάγη και μάλιστα θα έλεγα ότι θα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των εμπειρογνωμόνων εδώ ε, πάντοτε είμαστε ευτυχείς όταν ερχόμαστε στις Βρυξέλλες και όταν θέλουμε να έχουμε επαφή με τα θεσμικά όργανα και την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Άλλο ένα θέμα ήταν το ερώτημα των σχέσεων που έχουμε με την ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Επιτροπής αλλά και τις άλλες διευθύνσεις. Κοιτάξτε να δείτε, το 7ο πρόγραμμα για το περιβάλλον δεν είναι μόνο πρόγραμμα δράσης για την έμφυλη κλίμα, είναι ένα πρόγραμμα δράσης για όλα τα θεσμικά όργανα. Άρα λοιπόν προφανώς έχουμε και εμείς επαφή με πολλές άλλες επιτροπές, γενικές διευθύνσεις, Και ε, είναι προφανές ότι τα προγράμματα παραγωγής και κατανάλωσης δεν είναι λογικά και δεν εντάσσονται στα πλαίσια του περατού μας πλανήτη. Οπότε προσπαθούμε ε, να εστιάσουμε την προσοχή στην βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση στα θέματα ενέργειας, τροφίμων, ε, γεωργίας και άλλα και έτσι να συμβάλλουμε στη συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες για το θέμα της εφαρμογής και το θέμα των ευρωπαϊκών ελέγχων επιθεωρήσεων, εδώ θα ήθελα να είμαι πολύ προσεκτικός. Το DNA του οργανισμού μας είναι ότι δεν προβαίνουμε εμείς σε επιθεωρήσεις, ελέγχους. Αυτό θα άλλαζε τη σχέση που έχουμε με τους ε, τέρους IONET. Ριζικά Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο εμπιστοσύνης, ανταλλαγή σε στοιχείων, ανοιχτό σε κάθε είδους ε, στοιχεία ε, με εξασφάλιση και εμπιστοσύνη. Εάν τώρα αρχίσουμε και έχουμε εμείς ε, ρόλο επιθεώρηση ελέγχου, θα αλλάξει τελείως ο ρόλος που είχαμε μέχρι τώρα και σίγουρα δεν είμαστε υπέρ. τα στοιχεία που δίνουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτού του είδους τη λειτουργία από άλλους. Ναι, μάλλον και είμαι βέβαιος γι' αυτό και τα τελευταία πέντε χρόνια και πάλι ασχολούμαστε με εργασία αξιολόγησης πολιτικής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους ώστε να, κάνει εργασία, να κάνουν εργασία πιο κοντά στην εφαρμογή στην υλοποίηση. Για την απόδοση των ε, πόρων έχουμε συντάξει, έχουμε καταρτήσει μάλλον δείκτες, συνεργαζόμαστε και με τον ΩΣΑ και με την ΕΤΕΠ για τα θέματα αυτά, για το πώς δηλαδή επενδύουν ε, για τα στα προγράμματα αποδοτικότητας των πόρων, αν μπορούμε να επιταχύνουμε τις εξελίξεις Μακάρι να μπορούσα να πω ναι και να είμαι τόσο αισιόδοξο. Είναι προτεραιότητα για μας και το 2014 είναι αυτό προτεραιότητα και υπό το φως της πράσινης εβδομάδας και της εργασίας της Κομισιόν. Θέλουμε να στηρίξουμε τη δουλειά της Κομισιόν. Ταυτόχρονα, αν θέλουμε να, είμαστε, να έχουμε στέρεες πληροφορίες και στέρεους δείκτες που μας, προχω... που ε, Τροθούν ένα βήμα πιο πέρα οι επαφές με την νότιση και με το νόσα μας δείχνουν ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και από την άλλη πλευρά το να μην είμαστε ανοιχτοί σε βασικές επικρίσεις για την ποιότητα της εργασίας που κάνουμε ε, απαιτεί ότι πρέπει να ε, αφιερώσουμε κάποιο παραπανήσιο χρόνο. Ωστόσο, εστιάζουμε στην αποδοσή των πόρων και την αποδοτικότητα των πόρων. Ε, όπως στο έβδομο πρόγραμμα έτσι και θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε κάποια ε, σε ασχολίες μας αλλά για την Επιστημονική Επιτροπή θα έλεγα ότι είναι το αντίθετο συμβαίνει από την εντύπωση που έχετε. Μάλιστα, μόλις ολοκληρώσαμε μια εντατική εργασία, συνεργασία με την Επιστημονική μας Επιτροπή μέσω σεμιναρίων και δύο συναντήσεων που είχαμε μαζί τους, όπου προέκυψε ένα πενταετές πρόγραμμα εργασίας για την Επιστημονική Επιτροπή. Προχωρήσαμε δηλαδή, δεν είναι πια ad hoc προσέγγιση μας στην εργασία τους, έχουν ένα πενταετές πρόγραμμα συνδυασμένο με το δικό μας, όπου τα αναδυόμενα προβλήματα και τα θέματα βεβαιότητας και περιπλοκότητα είναι στο επίκεντρο των όσων εμείς θα κάνουμε. Είμαστε λοιπόν πλήρως ε, ε, δεσμευμένοι σε στρατηγική διαδικασία. Για το IONET κάναμε μόλις αναθεώρηση, κάναμε μια μεγάλη συνάντηση με τα εθνικά σημεία επαφής και εργαζόμαστε για αυξημένη αποδοτικότητα και συμμετοχή και ξέρω πως πρέπει να γίνουν κάποια βήματα εδώ. Αλλά αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα εργασίας που έχουμε ορίσει για το 2014 και της ε, μεγαλύτερης αποδοτικότητας. Το βασικό είναι ότι πρέπει να είναι αμφίδρομη η διαδικασία. Το IONET δεν μπορεί να είναι μόνο ένα δίκτυο που μας δίνει πληροφορίες, γιατί θα είναι μόνο μία διαδικασία παραγωγής στοιχείων, ενώ εμείς θέλουμε να είναι αμφίδρομη η διαδικασία και το 2015 θα είναι μια καλή ευκαιρία για να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και να ξεκινήσουμε ε, στενότερη συνεργασία και εδώ το δίκτυο, το AFP και το AONET θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για τα ερωτήματα του κυρίου Ζέμπερ. Ίσως κάπως προκλητικά να πω ότι κατάλαβα την ερώτησή σας ότι εννοεί ποια είναι η προστιθέμενη σας αξία στην διαδικασία ολόκληρη δηλαδή οικονομία, πράσινη ανάπτυξη κτλ. Να σας πω, καταρχήν ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Δουλεύουμε για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, τη βιωσιμότητα. Αυτά είναι τα θέματα για τα οποία δουλεύουμε. Επίσης, πολύ, πολύ κοντά στο ε, κεκτημένο δουλεύουμε. Ε, όσον αφορά το input για την παρακολούθηση της ε, εκθέσεις. Ε, κατ' ουσίαν επίσης ε, συνεργαζόμαστε με την Eurostat, τον ΟΣΑ και διάφορους άλλους διεθνείς οργανισμούς και αυτή είναι η πρώτη μας σύνδεση με την ευρύτερη βάση γνώσεων. Επιπλέον όμως ο τρόπος με τον οποίο τώρα η Ευρώπη προσεγγίζει τις περιβαλλοντικές και τις κλιματικές ε, πολιτικές εξορισμού αφορά και ευρύτερα ζητήματα. Οπότε συμβάλλουμε και στηρίζουμε την Κομισιόν στο πώς να απαντήσει ας πούμε στη διαδικασία του εξαμήνου και εδώ είμαστε πολύ ε, κοντά στα όσα εσείς αναφέρατε. Ε, συνεργαζόμαστε με το γραφείο του επικεφαλής επιστήμονα της του Επιτρόπου Μπαρόζο, του πρόεδρου Μπαρόζο, με συγχωρείτε, Είμαστε δηλαδή πολύ πολύ κοντά στα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν, αλλά μέσα στο πλαίσιο των, της εντολής μας. Η συστημική προσέγγιση είναι κοινωνιακή και οικονομική, γιατί αγγίζει τα συστήματα ενέργειας, τα συστήματα παραγωγής, οπότε κινείται όλο και πιο κοντά σε, αυτήν την, σε αυτά τα θέματα. Τεχνολογική καινοτομία, πώς, αυτές, πώς αυτή λαμβάνεται υπόψη στην ε, ΣΟΕΡ εξετάζουμε την καινοτομία για συγκεκριμένα θέματα αλλά και το παγκόσμιο πλαίσιο εκεί όπου αυτό συμβαίνει είναι βασική εργασία του ΣΟΕΡ ώστε να δούμε πώς τα στοιχεία μας εντάσσονται μέσα στην ε, ε, προοπτική της ανάλυσής μας και αυτού του είδους της εργασίας. Για τα φαρμακευτικά, το νερό και τη σχέση με την υγεία. Αυτά λαμβάνονται υπόψη στο τομέα που εργασίας υγεία και περιβάλλον, που είναι η ευρύτερη πλατφόρμα που αφορά αυτό το θέμα και πάλι σε σχέση με τα όσα είπε ο κ. Το κάνουμε αυτό με την Επιστημονική Επιτροπή αλλά και με άλλους. Μεταξύ αυτών είναι οι επιτροπές που ε, σας απασχολούν εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και οι οργανισμοί επίσης που σας απασχολούν εδώ. Επίσης ε, το κάνουμε σε συμφωνία με τους κανονισμούς και τις οδηγίες για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι να παρακολουθούμε. Δηλαδή τα στοιχεία που έρχονται είναι τα στοιχεία που είναι ήδη εντός του κεκτημένου. Αν το κεκτημένο περιλαμβάνει τέτοιου είδους στοιχεία, τότε πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Για να απαντήσω στον κύριο Ντέιβις και τις δικές του παρατηρήσεις, αν η Κομισιόν εισακούει την οργανισμό και αν έχουμε αντίκτυπο ή επηρεάζουμε. Θα έλεγα ότι αυτό εξαρτάται από διάφορα στοιχεία. Καταρχήν, και αυτή είναι και η βάση των όσων κάνουμε, είναι η ποιότητα της δουλειάς μας. Αυτή είναι η πρώτη μας ευθύνη. Εάν δεν μπορούμε να φτιάξουμε ε, πληροφορίες ε, ποιότητας ε, ευανάγνωστης και έβλεπτης, τότε δεν θα μπορέσουμε και να επηρεάσουμε και τόσο πολύ. Δεύτερον, συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν και ιδιαίτερα τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλίματος, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα ποιε κοινέ διαδικασίες θα μας βοηθήσουν ώστε να έχουμε στοιχεία για να βοηθήσουμε στις διαδικασίες ε, σχηματισμού πολιτικής. Ας πούμε, το, η δουλειά που κάναμε για το, την ποιότητα του αέρα στα αστικά κέντρα είναι ένα καλό παράδειγμα. Η εργασία που κάνουμε για να στηρίξουμε την διεύθυνση κλίματος με τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το UFCCC είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα. Τώρα, το πότε θα έχουμε... Όποτε έχουμε ποιοτικές πληροφορίες λοιπόν, προσπαθούμε να στηρίξουμε την ε, Κομισιόν και προσπαθούμε επίσης ε, να συμμορφωνόμαστε με την ε, ατζέντα κάθε φορά της Κομισιόν. Στις 9,5 μήνες που είμαι σε αυτή τη θέση έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις με την Κομισιόν για να τη συζητήσουμε αυτή την ατζέντα και πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε και θα έλεγα ότι η επιρροή μας είναι υπαρκτή. Αλλά εγώ το βλέπω όσοι εξή έχουμε μια κάποια ανεξαρτησία για το πώς προσεγγίζουμε τα πράγματα. Αλλά το τι κάνουμε θα πρέπει να συνδυάζεται και με την ατζέντα της πολιτικής εδώ στις Βρυξέλλες. Νομίζω πως είμαστε στο σωστό δρόμο λοιπόν και για διάφορα θέματα η επιρροή μας είναι μάλλον ψηλότερη από ό,τι θα πίστευε κανείς. Τελευταία ερώτηση είναι κατά πόσο πιστεύετε ότι θα υπάρξουν πολλές, πολλές, πολλοί επιπλέον κανονισμοί, αν χρειάζονται επιπλέον κανονισμοί. Καταρχήν ο ρόλος της υπηρεσίας δεν είναι να φτιάχνει κανονισμούς όπως ξέρετε. Ούτε στρέφεται κανείς εμάς για να μας ρωτήσει αυτή την ερώτηση, κανονικά. Εγώ πιστεύω πως μπορούμε να στηρίξουμε την ατζέντα περί αριθμίσεων ε, με διάφορους τρόπους. Αν δείτε ας πούμε που βρισκόμαστε με το έδαφος για την ώρα. Δεν παρεμβαίνουμε στη διαδικασία, αλλά τονίζουμε νέα ε, χρήση του εδάφους, ε, της γης, της κατά... και αυτό λόγω της προσαρμογής στο κλίμα ε, και αυτή η εργασία θα στηρίξει μια νέα αριθμιστική ατζέντα για το θέμα αυτό των εδαφών, αλλά εμείς δεν πιέζουμε για αυτήν την ατζέντα, εμείς παρέχουμε μια βάση γνώσης ε, που μπορεί να βοηθήσει. Τώρα, αν υπάρχουν άλλες ανάγκες σε σχέση με κανονισμούς, νομίζω πως η συστημική μας ατζέντα στέλνει μηνύματα όσον αφορά τη συνοχή και το είδος του κανονισμού που μπορεί να απευθύνεται σε πιο συστημικά ζητήματα. Αλλά και πάλι μένουμε στο δικό μας ρόλο, δίνουμε πληροφορίες που μπορούν να στηρίξουν τους όσους ε, θεωρούν πως υπάρχουν ευκαιρίες για τις διάφορες ρυθμιστικές ατζέντε και αυτά έχω να πω για αυτή την ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα έχουμε ένα πρόβλημα, το σύνθες πρόβλημα του χρόνου. Έχουμε την κυρία Άουφια, τη Λουκούσεβα, ένα σωρό συναδέλφου στον κατάλογο και έχουμε ξεπεράσει ήδη κατά 15 λεπτά την ώρα ε, που προβλέπετε θα ήθελα όλοι να κάνουν μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Όχι να αρχίσουν να αναπτύσσουν θεωρίες, μία ερώτηση. Ένα λεπτό. Για να έχουν ε, την δυνατότητα όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Ο κύριος. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω. Κύριε Διευθυντά, απαντήσατε ήδη στην πρώτη μου ερώτηση για την εις βάθος παρακολούθηση. Δεν θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Χαίρομαι για το πενταετές πρόγραμμα εργασίας σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνδέσει την επιστήμη με την πολιτική της στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για την Βιοπικιλότητα. Και επίσης χάρη στην πρωτοβουλία, την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει ενεργά και στην διακυβερνητική επιστημονική πλατφόρμα για τη βιοπικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Πώς λοιπόν το ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος συνεργάζεται με αυτή την διακυβερνητική επιστημονική πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποδειγματικός ε, ο κύριος Πρόντι επόμενος. Ehm, Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την αναφορά σας στο Κοπέρνικο. Και την αναφορά που κάνατε στο έδαφος. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα για την προσαρμογή μας στις κλιματικές αλλαγές και θα πρέπει να προχωρήσει με ταχύς ρυθμούς, γιατί το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό της ε, βιωσιμότητας, της αηφορίας. Δεν νομίζω ότι λίγη πράσινη μπογιά θα μας, ε, και λίγες καλοπιστικές προσπάθειες ε, θα μας εξυπηρετήσουν. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία εδώ και όχι για τα υλικά αγαθά και όχι μόνο για τα υλικά αγαθά προς κατανάλωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κοινό καλό. Και νομίζω ότι είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος να δώσει σωστές συστάσεις για τα θέματα αυτά. Επόμενος ο κ. Κουκοβίτς. Η κυρία Κουκοβίτς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον ε, Διευθυντή για την πολύ εξαντλητική αυτή παρουσίαση. Ναι, ναι, ναι, θα περιμένω να βάλω τα ακουστικά σα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς. Κύριε Διευθυντά, ήταν πραγματικά πολύ διεξοδική η ενημέρωση που μας κάνετε και εμπεριστατωμένη. Έχω μια απλούστατη ερώτηση που απασχολεί όμως ε, πολλούς και αφορά τη μέρημνα για την ε, δημόσια υγεία, για την ανθρώπινη υγεία. Έχετε μελέτες επιπτώσεων για το πώς ε, η όλη πολιτική θα επηρεάσει και την οικονομική ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μιλούμε για το όραμά μας και την πολιτική μας μέχρι το 2050 σχεδόν. Έχετε κάποιες εκτιμήσεις για το πώς μπορούμε να παρασκευάσουμε υγιεινά τρόφιμα για δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόουζα. Η κυρία Σόουζα. Σουίτσα μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταπληκτική η παρουσίαση του προγράμματος δράσης για το περιβάλλον για την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ θερμά. Έχω μία ερώτηση για να περάσουμε από το γενικό στο ειδικό. Πώς ε, οι γνώσεις αυτές ε, που συγκεντρώνεται μπορούμε, μπορούν να εφαρμοστούν στην πρακτική. Εμένα με ανησυχεί και με προβληματίζει ιδιαίτερη κατάσταση στη θάλασσα, τη Μεσόγειο, την Αδριατική, τον Εύξενο Πόντο. Γιατί δεν είναι όλε οι χώρε που περιβρέχονται από τι θάλασσε αυτέ ε, μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα δεν εφαρμόζουν το κοινοτικό κεκτημένο. Πώ λοιπόν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο και πώ ε, η AONET μπορεί να στηριχθεί στην εμπιστοσύνη και όχι μόνο στου νόμου, γιατί εσεί δεν έχετε αρμοδιότητα για υποβολή νομοθετικών προτάσεων. Πώ μπορείτε λοιπόν να συμβάλλετε στην εναρμόνιση και στην ε, ένωση των πολιτικών ώστε να έχουμε μια εναρμονισμένη εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρένιξ, λέει ο κύριο Σέικχαουτ, έχω μια γενική ερώτηση, γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο και το έργο του. Την τελευταία όμω πενταετία, Ποιε ήταν ε, οι πιο δύσκολε συζητήσει που είχαμε στι Βρυξέλλε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, συνήθω, για να μην πω συχνά, είναι τα όργανα πολιτική όταν λέμε αν θέλουμε μετά το 2021 έναν ή τρεις στόχους. Τι θα κάνουμε με, το, με τα βιοκαύσιμα, τι θα κάνουμε με τα ποσοστά πίσας, με την ε, σύστημα εμπορίας εκπομπών. Όλα αυτά είναι εργαλεία πολιτικής. Και όταν είπατε να μην εγκλωβιστούμε στην τρόχουσα κατάσταση, αλλά να είμαστε πιο διορατικοί, να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά τους σπόρους, να στηριζόμαστε στην βιοπικιλότητα. Το θέμα είναι με βάση τους ε, δείκτες ε, τι εργαλεία πολιτικής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποφύγουμε αυτόν τον εγκλωβισμό στην τρέχουσα κατάσταση και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ε, σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Λιούπτσεβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του ΕΟΠ για την πολύ χρήσιμη αυτή παρουσίαση που μας έκανε και που μας ε, ενημέρωσε για το πρόγραμμα δράσης ε, για το περιβάλλον του ΕΟΠ. Νομίζω ότι η πρόληψη των κινδύνων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα από ότι η εκ ε, αντίδραση και θεραπεία. Οπότε χρειαζόμαστε την εκτίμηση των κινδύνων το ίδιο με την παρακολούθηση της εξέλιξης κατάστασης. Έχετε όμως αρκετούς πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους για να ανταπεξέλθετε στην αποστολή σας. Γιατί όλα αυτά τα μοντέλα και τα δεδομένα που συγκεντρώνετε είναι πολύ σημαντικά για τα κράτη-μέλη για να προληφθούν οι κίνδυνοι και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, έχω και εγώ μια γενική ερώτηση, όπως και ένας προλαλής Ο ΕΟΠ πριν από ένα χρόνο εκπώνησε μια καταπληκτική έκθεση, το δεύτερο τόμο, με την αρχή της προφύλαξης και της καινοτομίας και κάποια πρόωρα σημάδια. Ε, πώς θα αξιοποιήσετε τα καταπληκτικά συμπεράσματα της έκθεσης εκείνης, κυρίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, που δυστυχώς εφαρμόζεται όλο και λιγότερο στην πράξη. Ευχαριστώ. Ήταν η τελευταία μιλητρία που είχαμε στον κατάλογο, οπότε δίνω το λόγο στον Διευθυντή του ΕΟΠ για σύντομες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ λακωνικός στις απαντήσεις, όπως ήταν επιγραμματικέ και ερωτήσει. Κύριος ο κύριος Φράγκο, ο πρώτος ε, ομιλητής στο δεύτερο γύρο. Θα ήθελα να πω ότι το έργο μας για την βιοπικιλότητα και τις υπηρεσίες λύση οικοσυστημάτων, για, τη, για τα λογιστικά σε ό,τι αφορά τις φυσικούς σπόρους και τα οικοσυστήματα. Ε, όλα αυτά ε, συγκεντρώνονται σε ένα σύστημα πληροφοριών της Ευρώπης και επίσης συνεργαζόμαστε στενά με τις παγκόσμιες πλατφόρμες. χθε ε, συναντήθηκα με εκπροσώπους της UNEP για να συμβάλλουμε και εμείς ως ΕΟΠ στο έργο των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα αυτά. Και έχουμε στενή συνεργασία και με άλλους φορείς, είτε είναι πιο ε, επιστημονική όπως είναι η πλατφόρμα TIP ή πιο μεθοδολογική ε, διαδικασία σαν αυτές της Νέας Υόρκης ή πλατφόρμες για παροχή δεδομένων όπως η UNEP ε, υπό την αιγύδα του γραφείου του Ναϊρόμπι. Φυσικά έχουμε στενή συνεργασία και θα συνεχίσουμε να έχουμε στενή συνεργασία με τους φορείς αυτούς. Κύριε Πρόντι, συγγνώμη καταρχήν που καθυστέρησα να βάλω τα ακουστικά μου για το Κοπέρνικο και τη χρήση εδάφους. Ε, ευχαριστώ και θα ήθελα να πω ότι το θέμα του εδάφους δεν περιορίζεται μόνο, στη, μόνο στο έδαφος, αλλά το έδαφος και οι ευκαιρίες που μας δίνει το Κοπέρνικος να μιλήσουμε για αλλαγή χρήσης γης και άλλα τέτοια συναφή θέματα είναι πολύ ενδιαφέρουσες ευκαιρίες και συμφωνώ για και θεωρώ ότι η προοπτική της μετάβασης που συμπεριλάβαμε στο πενταετές μας πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη και αυτό το στόχο, γιατί όταν μιλούμε για αλλαγές στην κοινωνία, Φυσικά περιλαμβάνουμε το πολιτιστικό κεφάλαιο, το ανθρώπινο κεφάλαιο και διάφορα άλλα στοιχεία. Όλα αυτά τα έχουμε υπόψη και σε συνεργασία και με άλλους φορείς προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε γνώση και να κάνουμε έργο αξιολόγηση ώστε να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα. Πάντως στον 20ο αιώνα είχαμε καλές επιδόσεις για πολλά θέματα αλλά δεν λάβαμε υπόψη τα όρια. Ενώ τον 21ο αιώνα Ελπίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα όρια. Και αυτή είναι πολύ σημαντική η μεταστροφή και στην νοοτροπία, αλλά και στην ε, χάραξη της πολιτικής. Και θέλουμε να συγκεντρώσουμε γνώσεις για να συμβάλλουμε με την παροχή τέτοιων πληροφοριών στους ηθήνοντες και όσους χαράζουν πολιτική. Κυρία Κουκόβιτς, φυσικά θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη το θέμα της υγείας και πιο ολοκληρωμένες μελέτες επιπτώσεων. Τώρα πώς συνδυάζεται αυτό με την οικονομική ανταγωνιστικότητα και το ε, πράσινο θεματολόγιο. Θα επικεντρωθούμε σε διάφορα θέματα. Καταρχήν, ε, είμαστε συνδεδεμένοι και με την διαδικασία του εξαμήνου. Οπότε έχουμε ήδη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Συνεργαζόμαστε και με άλλα θεσμικά όργανα για να παρέχω για να χορηγούμε γνώση ότι αφορά μια ουσιαστική πραγματική οικολογική οικονομία, πράσινη οικονομία. Και η ανταγωνιστικότητα στο μέλλον θα πρέπει να στηρίζεται και στις ε, προκλήσεις ε, της ε, οικονομίας με λίγο άνθρακα, λίγη χρυσή, χαμηλή χρυσή άνθρακα, ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και με τη λήψη υπόψη των ορίων γιατί μας ενδιαφέρει η οικολογική καινοτομία και σίγουρα η ανταγωνιστικότητα στο μέλλον θα περάσει και από αυτό το θέμα και θέλουμε να πρωτοστατούμε παγκοσμίω σε τέτοια ζητήματα. Εμείς στο ΝΕΟΠ θα δείξουμε πώς δείκτες της πράσινης οικονομίας εντάσσονται σε ένα πιο ανταγωνιστικό σύστημα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την εντολή μας. Δεν έχουμε τις αρμοδιότητες ούτε τις ικανότητες της Eurostat ή άλλων φορέων για πιο, για πιο μακροοικονομικούς ε, υπολογισμούς και προβλέψεις. Επίσης εξετάζουμε και κάποια οικονομικά εργαλεία όπως πράσινοι φόροι, οικολογικοί φόροι, συστήματα επιχορηγήσεων. Αυτά ανήκουν στα οικονομικά δημοσιονομικά εργαλεία για τη δημιουργία μιας ε, ανταγωνιστικής οικονομίας, αλλά θα πρέπει να είμαστε σεμνοί και μετριόφρον σε όλη αυτή τη συζήτηση. Η κυρία Σουίτσα. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη αυτή η γνώση. Εμείς ε, παρέχουμε γνώσεις και ελέγχουμε κατά πόσο εφαρμόζεται το κοινοτικό κεκτημένο. Στην πράξη και πώς, επηρεάζει, πώς επηρεάζεται το περιβάλλον και πώς επηρεάζονται και οι κάτοικοι της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον έλεγχο των ε, πολιτικών και για την ε, εξακρίβωση της υλοποίησης των στόχων που έχουμε θέσει. Οπότε σίγουρα η γνώση έχει έμπρακτη εφαρμογή εφαρμόζεται εμπράκτος και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όσοι ε, εργάζονται σε εθνικό επίπεδο και οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση. Τώρα, ρωτήσατε κάτι για τις θάλασσες. Μου άρεσε πολύ η ερώτησή σας, γιατί πριν από μια μισή εβδομάδα είχαμε, ε, μια, συμμετοχή σε μια διάσκεψη και στείλαμε εκθέσεις ε, για το θαλάσσιο περιβάλλον θα συνεχίσουμε τις αξιολογήσεις ε, των θαλασσών και ωκεανών και στην Ευρώπη και μάλιστα συνεργαζόμαστε με την ε, Σύμβαση για τον Εύξηνο Πόντο εν ώψη του ορίζοντα 2020 ε, με τη Συνθήκη για τη Μεσόγειο, για την Κασπία και θέλουμε με, τις, με τους εταίρους μας στην Ανατολή και στο Νότο εξετάζουμε με τις χώρες του Ευξήνου Πόντου και της Μεσογείου την κατάσταση στις θάλασσες αυτές. Εμείς ε, προσφέρουμε μια πλατφόρμα γνώσης για να στηριχθούν οι πολιτικές εκεί. Αλλά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πρόγραμμα για την προστασία της θάλασσας. Κύριε Έκχοτ, φαντάζομαι ότι οι συζητήσεις για τα εργαλεία της πολιτικής βρίσκονται στο επίκεντρο και μάλιστα στην προηγούμενη μου σταδιοδρομία που ήμουν επιστήμονας για θέματα πολιτικής, ε, με αυτό το θέμα μου κυρίως. Και το έργο του ΕΟΠ, ακριβώς για την αξιολόγηση των πολιτικών, αναφέρεται και σε εργαλεία και στο πώς ε, εφαρμόστηκαν και λειτουργήσαν τα εργαλεία. Το έργο για τους οικολογικούς φόρους, για παράδειγμα. Το έργο μας για τις επιδοτήσεις οι αξιολογήσει όλων αυτών των θεμάτων εντάσσονται σε αυτή την προοπτική. Και επίσης ε, έχουμε ένα πρόγραμμα αξιολόγηση των πολιτικών σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή πολιτική και αυτή είναι μια πολύ σκεμμένη επιλογή. Γιατί είναι η άλλη όψη του νομίσματο. Αν αποφασίσετε να επικεντρωθείτε περισσότερο σε εφαρμογή των πολιτικών, η αξιολόγηση της πολιτικής είναι σημαντικό ψηφιδωτό της όλης πολιτικής και ψηφίδα μάλλον του ψηφιδωτού της πολιτικής και θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση και των εργαλείων για να δούμε πώς εφαρμόζεται μια πολιτική. Και με το έργο μας ε, εξυπηρετούμε και αυτό το στόχο και συμβάλλουμε σε όσους ε, εφαρμόζουν τις πολιτικές. Με ρωτήσατε αν ε, είναι επαρκείς οι δείκτες που εκπονούμε. Σε όσους μας αποκαλούν Ινστιτούτο ε, δικτών και δεδομένων, εμείς λέμε ότι είμαστε Ινστιτούτο Γνώσης, Οργανισμός Γνώσης. Φυσικά χρειαζόμαστε δείκτες, αλλά για να παράγουμε γνώση, όχι απλώς ε, θόρυβο, ε, φασαρία δηλαδή και καταιγισμό πληροφοριών. Η γνώση είναι το ζητούμενο σε τελική ανάλυση. Και τελευταίες δύο ερωτήσεις, κύριε Λιπτσεβα Μάλλον έχω κατακρεουργήσει το όνομά σας στην προφορά. Κύριε Λιούπτσεβα, αρχή προφύλαξης ε, και πρόληψη των κινδύνων. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς θεωρούμε την πρόληψη των κινδύνων ε, βασικό στοιχείο της ε, χάραξης πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατοχυρώνεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και, και στο παρελθόν αλλά και στη συνέχεια θα συμβάλλουμε στην αναγνώριση της, των κινδύνων ώστε να συμβάλλουμε στην πρόληψη. Έχουμε μεθόδους για κάτι τέτοιο. Τώρα για τις σπόρους έχουμε στενή συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή και με άλλους φορείς της γνώσης, αλλά συνεργαζόμαστε και με το JRC, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, γιατί εκεί έχουν πολύ περισσότερα μοντέλα και ικανότητα για, δημιουργία μοντέλων. Εμείς δεν έχουμε τέτοια, τέτοιες δυνατότητες. Οπότε έχουμε συνεργασία και με αυτό το, το, τον φορέα. Τελευταία ερώτηση. Ναι, φυσικά χρειάζεται η αρχή της προφύλαξης και την ε, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη γιατί είναι από τις ε, θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος. Και μάλιστα θα διοργανώσουμε μια διάσκεψη για ανταλλαγή ιδεών στις Βρυξέλλες ώστε να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος και να μην παρελθοντολογούμε, αλλά να αξιοποιήσουμε το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα και να το εφαρμόσουμε στο μέλλον γιατί έχουμε μακροχρόνιους ορίζοντες 2020, 2030, 2050 και θα πρέπει για τις περιόδους αυτές να δούμε τι σημαίνει αβεβαιότητα και πώς θα, δούμε, θα αντιμετωπίσουμε την πρόληψη των κινδύνων. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπράουνιξ για την ε, ενδελεχέστατη απάντηση των ε, ερωτήσεων. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας σας και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία με την Επιτροπή περιβάλλοντος. Είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα κάνουν και οι επόμενοι συνάδελφοι της επόμενης επιτροπής, γιατί εδώ ολοκληρώνουν τις δικές μας εργασίες για την τρέχουσα θητεία. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα των νέων τροφίμων. Εδώ η συγητής είναι ο James Nicholson, ο οποίος και παίρνει το λόγο πρώτος. Ο κύριο Νίκολσον λοιπόν έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Θα θυμάστε στις 18 Δεκεμβρίου πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία αναμενόμενη, πολύ αναμενόμενη πρόταση σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα. Και η μεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής θα θυμάται την προηγούμενη απόπειρα να αναθεωρηθούν οι, κανόνε για τα νέα τρόφιμα από το Μάρτιο του 2011 όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν μπόρεσαν να καταλήξουν στο Σύμφωνο τα πλαίσια συνδιαλλαγής τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαχώρισε τότε την κλωνοποίηση από τα νέα τρόφιμα και παρουσίασε ένα ξεχωριστό πακέτο για την κλωνοποίηση τον περασμένο Δεκέμβριο. Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ουσιαστικά ε, συνεχίζει από το σημείο που σταμάτησε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2011 και συμπεριλαμβάνονται πολλά στοιχεία τα οποία είχαν προτείνει ο εισηγητής και εσκιώδης Ο βασικός στόχος ό,τι αφορά την πρόταση για τα νέα τρόφιμα είναι, εξ όσων καταλαβαίνω, να αντικαταστήσει το τρέχον σύστημα αμοιβαίας κατανόησης με ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, γενικής και κεντρικής ε, με μια ιστορία και ένα ιστορικό μάλλον και ασφαλών χρήσεων από τρίτες χώρες και να δημιουργήσει έναν κοινοτικό κατάλογο ε, πιστοποιημένων νέων τροφίμων σύμφωνα και με τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξέλιξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μια διαδικασία σε ό,τι αφορά την ε, εκτίμηση του κινδύνου σε μια διαδικασία η οποία προκαλεί μεγάλη αγανάκτηση και ανησυχία και από τους καταναλωτές και από την ε, βιομηχανία. Ελπίζω με το Συμβούλιο να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα κανονισμό που θα είναι και κατάλληλος αλλά θα απαντήσει και στις ανησυχίες του κλάδου για τις μελλοντικές εξέλιξεις. Όπως είπα, πιστεύω ότι πολλά μεγάλα ζητήματα ήδη είχαν απαντηθεί και επιληθεί στην προηγούμενη διαδικασία το 2011 και η διαδικασία συνδιαλλαγής δεν σημαίνει ότι φυσικά μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και να πάμε σπίτια μας τώρα. Θα πρέπει να χθενήσουμε την πρόταση του 2011 και θα πρέπει να φροντίσουμε ότι δεν θα έχει μείνει ούτε ένα στοιχείο αδιευκρίνηστο. Μετά τις εκλογές θα ε, ολοκληρωθεί η πρόταση και δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα πάει το χρονοδιάγραμμα. Να σας δώσω όμως μια εκτίμηση σήμερα από την τελεγή απόψε. Και αν επανεκλεγώ, το οποίο εξαρτάται από το εκλογικό μου κοινό, τον Ιούνιο και Ιούλιο θα ήθελα να αποστείλω το κείμενο ε, προς μετάφραση, ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο και μέσα Σεπτεμβρίου προθεσμία για τροπολογίες τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο να ψηφίσει στην Επιτροπή και ελπίζουμε να υπάρχει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Φυσικά όλα αυτά είναι υποκειμενικά και αρκετά φιλόδοξα, αλλά είναι ο στόχος μας. Η μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2008 με την υποστήριξη των σκιωδών μας ζήτησα από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να διεξαγάγουν μελετή αντικτύπου προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα παραμεληθούν οποιοδήποτε παράγοντες σε ό,τι αφορά και την παλιά μελέτη αντικτύπου. Να ευχαριστήσω τους συντονίστες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το πολύ θετική αυτή η κίνηση. Ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτό κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών. Ελπίζω ότι η και πιστεύω ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να είναι μια πλατφόρμα για την καινοτομία και με όλα αυτά λοιπόν στην έκθεσή μου θα επικεντρωθώ σε τρεις βασικές ε, πτυχές. Τα βασικά κριτήρια για την εκτίμηση των νέων τροφίμων καταρχάς. Ο νέος χαρακτήρας λοιπόν παραμένει και παραμένει ουσιαστικά ε, στα επίπεδα του 1997. Τα κράτη-μέλη έχουν διαθέσει μια ρεαλιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εκτίμηση και την αξιολόγηση του τι αποτελεί νέο τρόφιμο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να οριστεί το νέο τρόφιμο προκειμένου να υπάρχει νομική βεβαιότητα για τον ε, κλάδο σε ό,τι αφορά την αφαίρεση κάποιων κατηγοριών και κάποιων ορισμών. Αυτό θα οδηγήσει σε νομική αβεβαιότητα. Σε ό,τι αφορά τις πράξεις κάθε εξουσιοδότηση, αυτό συνδέεται με το πρώτο μου σημείο σε ό,τι αφορά τις εξουσίες που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ορισμούς. Θα πρέπει να ασφαλίσουμε ότι ο δίκτυπος στον κλάδο οποιαδήποτε δευτερογενούς ε, νομοθεσίας θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μην αλλάζει ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού πέρα από αυτά που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο ρόλος των κρατών μελών. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, οικοδομήσει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη, ιδιαίτερα στην κατάταξη των νέων τροφίμων και στην παροχή των ε, φορέων του κλάδου σε ό,τι αφορά για τα νέα τρόφιμα. Θεωρώ ότι μπορούν να ακολουθήσουν λοιπόν τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές τη ΕΦΣΑ και αυτό ισχύει ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του κλάδου. Τελευταίο παράδειγμα, δυνατότητα συμπερίληψη μιας ενός καταλόγου με τα απορριφθέντα προϊόντα με σημαντικέ πληροφορίες σε ό,τι αφορά απορριφθεί στις εφαρμογές τέτοιων τροφίμων και από τρίτες χώρες και να περιλαμβάνονται και αρχές και διαφορετικοί τέτοιοι φορείς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η πρόσβαση στην αγορά και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε με την πρόταση αυτή τη λειτουργία της αγοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω και στα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και να ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση. Η κυρία Αγιούζο, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι για την εκ μέρους του ΕΛΚ για μια Ακόμη φορά επαναρχόμαστε στο θέμα των νέων τροφίμων μετά το 2010 που απορρίφθηκε η πρόταση. Τελικά δεν συμφωνήσαμε για τα κλωροποιημένα τρόφιμα με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Νίκολσον για την ε, συνάντηση που είχαμε τις προάλλες και εκεί κάναμε έναν απολογισμό της κατάστασης ε, και συμφωνήσαμε το Σεπτέμβριο κατά πάσα πιθανότητα να οργανώσουμε δημόσια ακρόαση για αυτό αυτή την πολύ σημαντική ε, νομοθετική πρόταση. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο κείμενο το νομοθετικό που είναι πιο σαφές ε, και συνάδει περισσότερο με την κοινή θέση του 2010. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι πολύ πιο εύκολη η διεκπαιρέωση νομοθετικής διαδικασίας με τη νέα πρόταση. Αυτό που με απασχολεί είναι το άρθρο 1 και ελπίζω να διασκεδαστεί αυτή η ανησυχία μου. Το άρθρο 1 λοιπόν αναφέρεται στην ε, η εισαγωγή στην αγορά των κλωνοποιημένων ζώων με βάση την οδηγία την επόμενη. Από τη στιγμή που συζητάτε όμως ε, οδηγία, τι να σας πω, εμείς δεν έχουμε ορίσει καν εισηγητές. Οπότε αν καθυστερήσει η έγκριση του κανονισμού, ίσως ε, αντιμετωπίσουμε και μία περίοδο νομικού κενού. Αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τους ορισμούς των νέων τροφίμων. Ο κύριος Νίκολσον, ο εισηγητής μας, αναφέρθηκε στον ορισμό που είναι ίδιος με αυτόν της πρώτης πρότασης. Και αναφέρεται σε τρόφιμα που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό πριν το Μάιο του 1997. Τι θα πει αυτό όμως, δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αυτά τα τρόφιμα Εβραίος πριν από το Μάιο του 1997. Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Επίσης μιλούμε για εύλογους ε, ε, παράγοντες ε, ή θεμητούς. Ποιοι είναι αυτοί οι εύλογοι ή θεμητοί παράγοντες ή θα πρέπει να τους ορίσουμε ή το να τους αφήσουμε σε, σε μεταγενέστερη κατεξουδότηση πράξη. Κάπως πάντως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν, είμαστε, δεν βλέπουμε και πολύ καλό μάτι της κατεξουδότησης πράξης και πολύ λιγότερο τις εκτελεστικές πράξεις, γιατί πολύ συχνά με τέτοιες πράξεις αλλάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αισθητά μία νομοθεσία που έχουμε ήδη ε, εγκρίνει. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά εξουδότηση πράξης ως εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τροποποιεί νομοθετικές ε, προτάσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Νίκολσον για τα απορριφθέντα τρόφιμα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Επίσης θα ήθελα να μου διευκρινίσει δύο σημεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα, και ένα θέμα που αφορά και τα απορριφθέντα τρόφιμα. Καταρχήν ε, για τα έντομα. Πολλές ερωτήσεις ε, έχω λάβει και μου τηλεφωνούν πολύ συχνά. Φαντάζομαι το ίδιο θα αντιμετωπίζει και ο εισηγητής. Αν απορριφθεί ότι ένα έντομο έχει επιστηστικό ιστορικό τουλάχιστον 25 ετών σε μια χώρα, θα πρέπει να θεωρηθεί νέο τρόφιμο ένα έντομο ή αν θα μπορεί να απορριφθεί η συμπερίληψή του στον κατάλογο για άλλους, στόχους που δεν θα είναι, λόγους που δεν θα είναι λόγια επισητιστικής ασφάλειας. Επίσης, ε, οι άδειε θα είναι γενικές ε, και απεριόριστες χρονικά, ενώ προβλέπονται προσωρινές ε, μεμονωμένες ατομικές άδειε πενταετούς διάρκειας σε περίπτωση που υπάρχει προστασία δεδομένων. Δεδομένου όμως ότι οι αποφάσεις για διοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα, θα απευθύνονται στον ετούντα την, άδεια εμπορευματοποίησης, θέσης εμπορία, ίσως δημιουργήσουμε διακριτική μεταχείριση με τη μεταφορά των πιο πρόσφατων αδειών ε, στο νέο κατάλογο. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια ειδική περίοδο για τα εγκεκριμένα τρόφιμα που δεν έχουν κοινοποιηθεί με βάση το άρθρο 4, 5 ή 7 του τρέχοντος κανονισμού, του 258 97 δηλαδή ή να περιληφθούν σε έναν ενιαίο κατάλογο για να μπορούμε να συγκρίνουμε αυτά τα τρόφιμα με αυτά που έχουν εγκριθεί με βάση το νέο κανονισμό και να έχουμε πενταετή περίοδο ε, σε περίπτωση που ισχύει η προστασία δεδομένων. Ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε ένα μεταβατικό μέτρο, μια μεταβατική περίοδο για τέτοιες περιπτώσεις. Κάτω του λοιπού, συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να εγκριθεί ο κανονισμός γιατί είναι πολύ σημαντικός και για τους καταναλωτές αλλά και για τη βιομηχανία και κυρίως για την τεχνολογική καινοτομία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Για τους φιλελεύθερους, επειδή έχουν ήδη διορίζει την Κορίν Λεπάζ ε, συντονίστρια και μετά έχουμε την κατήκα Λιωτάρ. Σας παρακαλώ όμως, ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα, αλλά σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας, γιατί δάλλως δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, ρόλο των ε, εθνικών οργανισμών. Στην πρόταση που μας υποβάλλεται, οι εθνικοί οργανισμοί έχουν τελείως ε, εξαφανιστεί. Ωστόσο, έχουμε διάφορα παραδείγματα που δείχνουν ότι οι εθνικοί οργανισμοί μπορεί να έχουν αποκλίνουσες απόψεις ε, με την ΕΦΣΑ. Χωρίς να αμφισβητήσουμε το κεντρικό ρόλο της ΕΦΣΑ, και θα μπορούσαμε, θα πρέπει να δούμε, ότι, να μεριμνήσουμε ότι θα υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι στο κείμενο. Δεύτερον, καταλάβαμε ότι η κλωνοποίηση δεν, ήταν δεν είναι πλέον το βασικό θέμα, ωστόσο ξέρουμε ε, σε αυτό το κείμενο, ωστόσο ξέρουμε ότι μια συγκεκριμένη νομοθεσία θα πάρει χρόνο. Οπότε, για αυτή τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να προβλέπετε από το κίνητο ότι η θέση στην αγορά κλωνοποιημένου κρέατος ή κρέατος μάλλον από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους, θα ρυθμίζεται ή θα, η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη και το πιθανό περιβαλλοντικό αντίκτυπο των νέων τροφίμων και μιλώ κυρίως για τις νανοτεχνολογίες. Και τέλος, τελευταίο σημείο για την εμπιστευτικότητα. Ε, χρειάζεται καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των δεδομένων των βιομηχάνων και την ενημέρωση του κοινού. Η σύμβαση Λαρούση απαιτεί ε, αρχούς συγγνώμη, ε, απαιτεί την ενημέρωση. Μπορούμε να κατανοήσουμε τον απόρριτο χαρακτήρα των βιομηχανικών στοιχείων, αλλά ό,τι έχει να κάνει με το αντίκτυπο στο περιβάλλον την υγεία είναι δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος και άρα θα πρέπει να δημοσιοποιείται. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τελευταία η καλή Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την συνάντηση την οποία διοργανώσαμε. Πραγματικά ήταν ωφέλιμη. Ήμουν η προηγούμενη εισηγητρία για το θέμα των νέων τροφίμων. Τότε δυστυχώς τη συνδιαλλαγή δεν τα βγάλαμε πέρα και θα ήθελα να αναφέρω γιατί δεν καταφέραμε να βγάλουμε αποτέλεσμα την προηγούμενη φορά, γιατί ουσιαστικά υπήρχαν δύο λόγοι, δύο λόγοι για τους οποίους δεν πετύχαμε αποτέλεσμα. Η κλωνοποίηση των ζώων για τρόφιμα, καταρχάς, γιατί το Κοινοβούλιο συμφωνούσε ότι θα έπρεπε να απαγορευτεί τότε η κλωνοποίηση ζώων για τρόφιμα και η εισαγωγή ε, ζωικών προϊόντων και σε ό,τι αφορά και τους απογόνους γιατί το Συμβούλιο δεν ήθελε καν να υπάρξει επισήμανση, να μην ξέρει να ρωτήσει για του απογόνου τέτοιων ζώων. Δεν συμφωνήσαμε λοιπόν και η συζήτηση συνεχίστηκε σε ό,τι αφορά την εμπορία προϊόντων, τροφίμων, αποκλοπημένα ζώα. Αυτό το θέμα λοιπόν έπρεπε να συνεχίσει να το επεξεργάζεται η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή μας. Ο δεύτερος λόγος τον οποίο δεν ολοκληρώθηκε στην διαλλαγή και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για όλες τις πολιτικές ομάδες, ήταν η κατεξουσιοδότηση πράξης. Πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κατάλογος των εγκεκριμένων νέων τροφίμων να ενημερώνεται με implementing acts, με εκτελεστικέ πράξεις. Το Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι αυτός ο κατάλογος ήταν ο πυρήνας της πρότασης της νομοθεσίας για τα νέα τρόφιμα και ως εκ τούτου επιμείναμε να είναι πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το ξέρουμε, είναι ένα οριζόντιο θέμα άλλωστε σε όλο το κοινοβούλιο, το οποίο ανακύπτει σε πάρα πολλέ ε, εκθέσει. Προτείνονται εκτελεστικέ πράξει, ενώ το κοινοβούλιο θέλει πράξει κατά Αυτό που με προκαλεί την πιο μεγάλη έκπληξη στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα νέα τρόφιμα, για τη νέα, επιτροπή, για τη νέα πρόταση, είναι ότι δεν ελευθεί καθόλου υπόψη ε, αυτή η στάση του Κοινοβουλίου στα άρθρα 7, 8 και 11 πάλι implementing acts, πάλι εκτελεστικές πράξεις προτείνουν. Αυτό μου φαίνεται χαζό από πλευρά ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε να επιδείξει κάποια πολιτική ευστροφία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό, γιατί ουσιαστικά το Κοινοβούλιο είχε συμφωνήσει με το Συμβούλιο σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Ε, άρα, καλό θα ήταν να έχει γίνει τώρα μία πρόταση όπου θα είχαν επανέλθει όλα τα στοιχεία από τα οποία είχαμε συμφωνήσει τότε με το Συμβούλιο και το πρόβλημα με τις εκτελεστικές πράξεις και τις πράξεις καταξιοδότησης που είχαμε τότε κάπως να είχε λάβει υπόψη και τη στάση του Κοινοβουλίου, εν πάση περιπτώσει. Όχι όμως. Γάιδαρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξανά χτυπάει στο ίδιο εμπόδιο για δεύτερη φορά. Κρίμα. Πάλι δύο-τρία χρόνια μπορεί να πάρουν οι διαπραγματεύσει για να ξαναξεκινήσουμε συζητήσει για θέματα για τα οποία είχε συμφωνήσει ουσιαστικά τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η, το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο, τα νανοτρόφιμα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Μία άλλη ιδέα τώρα που έχει αλλάξει για τα νέα τρόφιμα από τρίτε χώρε και τότε είχε συμφωνήσει Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη σημερινή, η διαδικασία της πιστοποίησης θεωρώ ότι έχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Με άλλα λόγια, δεν προσεγγίσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε προσεγγίσει πιο πολύ τις ιδέες επί των οποίων είχαμε συμφωνήσει στη συνδιαλλαγή τότε και να είχαμε απαλύνει και κάπως την διαμάχη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πρότασης για τις ε, πράξεις κατεξουσιοδότησης. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτα. Ε, Ευχαριστώ. Ναι. Συγγνώμη, δεν άκουσα ότι με δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Γίνεται μια συζήτηση πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε να κάνουμε με την καινοτομία και το κατά πόσο θα επιτρέψουμε την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής και να καθησυχαστεί όσον αφορά ερωτήματα και ανησυχίες που θα μπορούσε να έχει. Ένα θέμα που έθεσε ήδη η Κορίν Λεπάζ και που θέλω να επανέλθω όμω είναι η σχέση με του εθνικού οργανισμού. Αν και θεωρώ πω είναι πολύ καλό να έχουμε μια κεντρική διαδικασία, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει η σχέση με του εθνικού οργανισμού και θα ήθελα να γνωρίζω εάν υπάρχουν δυνατότητε προσφυγή στου εθνικού οργανισμού ε, από τη στιγμή που θα υπήρχαν αποκλήσει απόψεων για ε, κάποια τρόφιμα νέα. Και έπειτα, ένα κράτος μέλος θα μπορούσε μεταβατικά επί τη βάση μιας αξιολόγησης ή με βάση κάποια νέα στοιχεία να περιορίσει ή να αναστείλει την κυκλοφορία ενός νέου τροφίμου στην επικράτειά του αν θεωρεί πως μπορεί να ε, επιφέρει αυτό κινδύνους για τον καταναλωτή. Τέλος, ε, υπάρχουν και τίθενται διάφορα ερωτήματα με βάση τα νέα τρόφιμα και μάλλον τις ουσίες που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες ή που χρησιμοποιούνται και στον τομέα της ιατρικής. Έτσι. Βλέπουμε ας πούμε την κινέζικη ιατρική που μπορεί όμως να θελήσουν να μπουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια διότι θα έχεραν ε, του στάτους των νέων τροφίμων. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να τα απαντήσουμε μάλλον αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Και τώρα λοιπόν έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Μποσέτσι. Συγγνώμη για το όνομα και το πώς τον προφέρω. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Μποσέτσι. Σας ευχαριστώ. Μπρίτσι είναι το επώνυμό μου. Εν Δυστυχώ, ε, ο διευθυντή έπρεπε να πάει σε άλλη συνεδρία, συζητώ συγγνώμη. Θα τον να πληρώσω εγώ. Χαίρομαι για τα σχόλια που ακούσαμε και στόχος της πρότασης είναι να γίνει μια πλατφόρμα για την καινοτομία στην Ευρώπη και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα των τροφίμων. Βέβαια, η ενίσχυση της καινοτομίας και η πρόθεση της καινοτομίας δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της ασφάλειας των τροφίμων. Γι' αυτό και βελτιώσαμε τον κανονισμό. Ε, ε προβλέπουμε νέα διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης και ταχύτερο σύστημα έγκρισης. Επίσης, ε, αναμειγνύει τα κράτη-μέλη στην όλη διαδικασία, γιατί τα ενημερώνει για τις ε, πιθανές εφαρμογές για τις δυνατές εφαρμογές και επίσης ε, τα κράτη-μέλη συμμετέχουν και στη διαδικασία αδειοδότησης μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Συμμετέχουν και στο συντονισμό, στα πλαίσια της ΕΦΣΑ, του, του ΕΦΣΑ μάλλον, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων, που συνεργάζεται με τους εθνικούς αντίστοιχους φορείς. Ε, αυτό συμβαίνει και με τα παραδοσιακά τρόφιμα, αν δηλαδή μια χώρα θέλει να θέσει το εμπόριο παραδοσιακό τρόφιμο, αν κανένα κράτος μέλος ή ο ΕΦΣΑ δεν ε, εκφράσουν αντιρρήσεις, ε, γίνεται δεκτή η κοινοποίηση. Στόχος λοιπόν δεν είναι να αποκλείσουμε τους εθνικούς οργανισμούς, ε, αλλά να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό που θα εξυπηρετεί και το στόχο της καινοτομίας αλλά και το στόχο της ασφάλειας των τροφίμων. Σε ό,τι αφορά την κλωνοποίηση, όπως ανέφεραν και ο συγγετής και κάποιοι, κάποια άλλα μέλη, αποκλείσαμε το θέμα της κλωνοποίησης γιατί έχουμε ξεχωριστό πακέτο για την κλωνοποίηση που θα τύχει ξεχωριστής επεξεργασίας και διαπραγμάτευσης. Φυσικά είναι πιθανόν οι προτάσεις για την κλωνοποίηση να μην εγκριθούν αρκετά γρήγορα ώστε να αποκλειστούν από τον κανονισμό αυτό τα ε, συνάφη τρόφιμα. Πάντως, ε, ίσως θα πρέπει να ε, προβλέψουμε μια διαδικασία προέγκρισης για τις αγορές για ε, προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα, ενώ όσο περιμένουμε την έγκριση της σχετικής οδηγίας για την κλωνοποίηση, για να αποφύγουμε κενό δικαίου. Επίσης θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση από τον παλιό στο νέο κανονισμό. Το σημαντικό είναι να αντιληφθούμε εδώ ότι σήμερα ακόμη και αν έχουμε ατομικές άδειες, είναι ατομικές αλλά μέχρι κάποιο ορίου, γιατί έχουμε μια επιπρόσθετη τεχνοκρατική διαδικασία. Δηλαδή, μετά την χορήγηση ατομικής άδειας σε, σε ένα παραγωγό νέου τροφίμου. Οποιοςδήποτε άλλος παραγωγός μπορεί να, να ζητήσει αντίστοιχη άδεια για ένα ισοδύναμο τέτοιου τροφίμου. Στην νέα πρόταση προβλέπουμε ότι αν μια εταιρεία έχει αναπτύξει καινοτόμα και επιστημονικά δεδομένα και με βάση τη δική της έρευνα παρασκεύασε ένα νέο τρόφιμο, δίνουμε την ευκαιρία σε αυτή την εταιρεία να θέσει το νέο τρόφιμο στην αγορά για μία πενταετία. Στην πενταετία αυτή θα είναι μόνη της η εταιρεία στην αγορά, εκτός για να επιτρέψει σε άλλες εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα της και τα επιστημονικά της ευρήματα. Θα είμαστε πάλι πολύ προσεκτικοί στην έμπρακτη εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης. Πάντως το κείμενο μας επιτρέπει κάτι τέτοιο για την ομαλή μετάβαση. Τώρα, στο κείμενο επιτρέπουμε παραδοσιακά προϊόντα ή γεωργικά προϊόντα να επωφεληθούν από το σύστημα κοινοποίηση. Και όπου επιτρέπεται τα συμπεριλαμβάνουμε σε έναν κοινοτικό κατάλογο. Το κείμενο της συνδιαλλαγής προτείνει χάριν σαφήνειας και για το συμφέρον των ε, επιχειρήσεων προτείνουμε ένα ενιαίο κατάλογο για όλα τα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα. Βέβαια μπορούμε να τα χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία προβλέπει εφαρμογή ε, για να μπει το τρόφιμα στον κατάλογο. Μετά έχουμε εφαρμογή περιορισμένης χρονικής διάρκειας, οπότε θα έχουμε το τρόφιμο αλλά με προθεσμία και τέλος άδεια που θα στηρίζεται στην κοινοποίηση. Εκεί επισημαίνεται ότι το τρόφιμο αυτό είναι αντικείμενο κοινοποίηση. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα θέση εμπορία γιατί η άδεια είναι γενική και οι φορείς μπορούν να παραπέμπουν σε ένα νέο κατάλογο. Είναι πολύ πιο εύκολο και για τις επιχειρήσεις αντί να χρειάζεται να ψάχνουν τις πληροφορίες σε πολλούς επιμέρους καταλόγους. Σε ό,τι αφορά τους ορισμούς, στη συνδιαλλαγή αποφασίσαμε να έχουμε έναν ορισμό που θα, θα παραπέμπει στην ε, ευρία κατανάλωση ενός τροφίμου από το 97 και μετά. Επίσης ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός οι κατηγορίες που υπάρχουν στον τρέχοντα κανονισμό μερικές φορές είναι παραπλανητικές. Για παράδειγμα τα έντομα. Έχουμε συζήτηση για το κατά πόσο τα έντομα εμπίπτουν στη μία ή την άλλη κατηγορία. Ενώ ο ε, του νομοθέτη τότε, στον προηγούμενο κανονισμό, το 1997, ήταν αν έντομα ή άλλα τρόφιμα δεν έχουν καταναλωθεί ευρέως, τότε θα πρέπει να θεωρούνται νέα τρόφιμα και να υπόκεινται σε αξιολόγηση της ασφάλειας. Επίσης, η αξιολόγηση της ασφάλειας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσκομα, ως ε, τροχοπέδι της ε, καινοτομίας, αλλά θα πρέπει η αξιολόγηση ασφάλειας να θεωρείται θετικό στοιχείο. Και είναι ένας ε, τρόπος η αξιολόγηση ασφάλειας για να κερδίσουν οι επιχειρήσεις την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και επίσης οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές θα εξασφαλίζουν ότι ένα νέο τρόφιμο που δεν έχει καταναλωθεί στο παρελθόν είναι ασφαλές και μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. Έχω την αίσθηση ότι απάντησα στις ερωτήσεις. Υπάρχει και το λεπτό θέμα των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Τα άρθρα που αναφέρονται σε εκτελεστικές πράξεις ε, πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει σχετική νομοθεσία. Οπότε πρόκειται για εκτελεστικές πράξεις ε, που αφορούν μη ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού. Άρα πληρείται ε, η προϋπόθεση για τις εκτελεστικές πράξεις. Αυτά νομίζω ότι απάντησα και ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή και τους υπόλοιπους ε, βουλευτές για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά τους. Ευελπιστώ ότι θα ολοκληρώσουμε το όλο θέμα στην πρώτη ανάγνωση. Σα ευχαριστώ. Θέλει και ο να πει δύο λόγια. Κλείνοντα, σα κύριε Νίκολσον. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι έχετε πίεση χρονική. Να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο και έκαναν ε, σχόλια, ιδιαίτερα τους ε, Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενους μήνες. Νομίζω ότι ενδεχομένω να εκφραστούν κάποιε ανησυχίε, ενδεχομένω να ανακύψουν κάποιε διαφωνίε και από το παρελθόν, αλλά από τον τρόπο που η συζήτηση σήμερα θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την ανησυχία τη κυρία Αγιούζο για τι πράξει κατά εξουσιοδότηση, ούτε εμένα μου αρέσουν και εγώ δυσκολεύομαι αλλά αυτό ισχύει και σε πολλούς άλλους ε, τομείς και σε πολλές άλλες εκθάσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ λοιπόν για τη συνεισφορά σας. Ελπίζω να είναι καλή η συνεργασία και να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό πριν από τα τέλη του Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νίκολσον. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτή η συζήτηση και το θέμα αυτό θα συνεχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε και μετά τις, με τις ευρωεκλογές. Ωραία. Και έτσι Φτάνουμε στο τελευταίο σημείο της μήνυσης διαταξής για σήμερα, στο 7 λοιπόν. Δημιουργία και λειτουργία ενός αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς για το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών. Σοφία Κονή. Επειδή έχει περάσει η ώρα να ζητήσω από όλους και από την εισηγήτρια να είναι σύντομη προκειμένου να Πάρε το λόγο, να πάρει το λόγο όλοι οι συνάδελφοι. Σοβή, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω τρένο στη 1 και 4, 1 και 13 για, για την ακρίβεια, οπότε και εγώ βιάζομαι. Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση της συζήτησης και της σκέψης ε, για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών. Και μετά την έκθεση Τελβό Σιμάνσκι για τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 Σήμερα ξεκινάμε την ανάλυση του νομοθετικού πακέτου του, της 22ης Ιανουαρίου με θέμα το αποθεματικό σταθερότητας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα είναι ο κρογωνιαίος λίθος της κλιματικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι ιδιαίτερος για την ευθύνη που μου αναθέσατε και θα συνεργαστώ με όλους για να βρούμε μια λύση προκειμένου να ενισχύσουμε και να σταθεροποιήσουμε αυτή την αγορά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ένα σημαντικό στοιχείο. Η ευρωπαϊκή αγορά άθρακα είναι μια τεχνητή αγορά που δημιουργήθηκε για πολιτικούς λόγους, γι' αυτό και θα πρέπει να ορίσουμε με πολιτικό τρόπο τους όρους λειτουργίας της, με συντονισμένο και βιώσιμο τρόπο. Οπότε η, ευρωπαϊκή αγορά, η δημιουργία της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα μοιάζει με την ε, εγκατάσταση παρκομέτρων σε μερικές κοινότητες σε μερικές περιπτώσεις είναι δωρεάν. Και το πάρκινγκ και η εκπομπή καυσαερίων. Αλλά ε, γίνεται επιπληρωμή προκειμένου να περιοριστούν οι δραστηριότητες αυτές και να περιοριστεί ο αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση είναι πολιτική. Η πολιτική αυτή απόφαση δημιουργεί μια αγορά που επαναλαμβάνω θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τεχνητή. Και η ιδιαιτερότητα του, της στάθμευσης επιπληρωμή είναι ότι οι τιμέ δεν είναι κειμενόμενε. ενώ η ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα είναι ότι η προσφορά ποσοστώσεων ε, καθορίζεται από μια πολιτική πολιετή απόφαση. Ε, η ζήτηση των ποσοστώσεων εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση και τις επενδύσεις που έχουν γίνει για τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων. Και σήμερα η αγορά αυτή ε, έχει μια πολύ χαμηλή τιμή, πολύ μικρή τιμή και μια διαφάνεια πολύ προβληματική γιατί οι επενδύσεις συνήθως έχουν μακροπρόθεσμο ή πολύ μακροπρόθεσμο προγραμματισμό ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. Εδώ το backloading και το πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 δίνει μια μερική απάντηση, υπερβολικά αποσπασματική και δεν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Η αγορά λοιπόν αυτή ε, υφίσταται το κίνδυνο της μεταβλητότητας των τιμών, η προσφορά είναι σταθερή αλλά οι τιμές κειμενόμενες και επίσης υπάρχει πρόβλημα που αφορά τη μετάβαση από την τρίτη στην τέταρτη φάση γιατί εκεί ίσως έχουμε μείωση των ποσοστώσεων μεταξύ 2020 και 2021. Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δύο δυσκολίες. Προτείνει καταρχήν τη δημιουργία ενός αποθεματικού σταθερότητας αγοράς που θα λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή θα περιορίζει τις διακοιμάνσεις ε, και προς τα πάνω και προς τα κάτω και μάλιστα από το 2021. Προτείνει επίσης την εφαρμογή μιας ε, ισορροπημένης μετάβασης μεταξύ των διαφόρων φάσεων. Δηλαδή θέτει ε, και εξορροπεί τις ποσοστώσεις για την τριετία 2020, ε, 2021 και 2022. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ουσιαστική συζήτηση, ψύχρεμη και χωρίς ε, συναισθηματισμούς για το θέμα αυτό. Και σίγουρα χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ε, ρύθμισης της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα τα θέματα είναι ανοιχτά και περιμένω τις προτάσεις. Τι μόρφη θα λάβει αυτή η ρύθμιση. Πολλές δυνατότητες. Αυτόματη διαχείριση των πλεονασμάτων ή έλλειψη ποσοστώσεων, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας των Ποσοστώσεων, με τη μορφή μιας ανεξάρτητης αρχής, ενός ανεξάρτητου φορέα. Και φυσικά είμαι ανοιχτή και περιμένω οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Το θέμα είναι, θα πρέπει να αποφύγουμε ή να εξασφαλίσουμε κρατικό έλεγχο, δημόσιο μάλλον έλεγχο του μηχανισμού αυτού. Άλλη ερώτηση. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να λειτουργεί σε αιτήσια βάση. Είναι καλή αυτή η λύση. Πώς θα τροφοδοτείτε το αποθεματικό. Ε, με τον νη 1 και με βάση τη χρονιά νη μείον 1. Μήπως έτσι επιβραδευτεί η διαδικασία και δημιουργηθεί μια αναλαστικότητα. Πώς θα αποφύγουμε τη μετατροπή του μηχανισμού αυτού σε ε, φενάκι ή σε αναποτελεσματικό μηχανισμό. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι στόχους θέλουμε να υλοποιήσουμε με την αυτή νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα την ασφάλεια δικαίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις μας στην τρίτη περίοδο, στην τρίτη φάση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να προβλέψουμε και μεταβατικό μηχανισμό για το τέλος της περίοδου. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα, ε, σαφήνεια του μηχανισμού, ε, γιατί η αγορά άνθρακα είναι ως λίθος, επαναλαμβάνω, της περιβαλλοντικής μας πολιτικής και τέλος, ε, κατά τη γνώμη μου, στόχος μας είναι να κάνουμε μια αντίστροφη συζήτηση από αυτή που κάναμε για το backloading. Μια ε, ψύχρεμη, ε, λογική συζήτηση χωρίς συναισθηματισμούς και πάθη για να βρούμε λύση ώστε η ευρωπαϊκή αγορά άθρακα να είναι βιώσιμη, πιο σταθερή και να αποτελέσει την τον πιο οικονομικό τρόπο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, συζήτηση, δεν έχουμε πολύ χρόνο για τη συζήτηση γιατί επίκειται και ευρωεκλογέ, αλλά τώρα ξεκινάει η συζήτηση που θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος και περιμένω, επαναλαμβάνω, τις απόψεις και προτάσεις σας. Συνάδελφε, ήμουνα ε, εισηγητή για το backloading και με είχε ρωτήσει τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι πότε θα συνεχίσαμε το backloading, μέχρι τα Χριστούγεννα, του 2012. Ρώτησα ποιο έτο εννοείται, τα Χριστούγεννα πιανού έτος. Ελπίζω εσείς να τα πάτε καλύτερα στην έκθεση αυτή, προκειμένου να πάνε καλύτερα τα πράγματα και λίγο πιο γρήγορα, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις. Ε, σήμερα το απόγευμα θα ληφθούν σημαντικέ ε, αποφάσει σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά κτλ. Ε, κατά πόσον το θέλουμε αυτό ή όχι, έχουμε μια επιλογή και θα δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα. Πέτερ Λίζε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για σήμερα το απόγευμα δεν θέλω να αποφανθώ ούτε να πάρω το λόγο να υποστηρίξω την Σοφή εικόνη στην ε, προσέγγιση της η οποία είναι ανοιχτή αλλά και επικοδομητική. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα πρόβλημα. Το backloading μας έχει δώσει λίγο χρόνο. Έχουμε πολλά πιστοποιητικά ε, και πάρα πολλά στο εμπόριο για τους ρηπούς. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα προς τα έξω, προς τον υπόλοιπο κόσμο, ότι είμαστε ε, σοβαροί και θέλουμε όντως να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος, να αποφύγουμε ακριβές λύσεις ε, αντί για μια ευρωπαϊκή λύση θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε το πνεύμα τη Σοφή Οκονή και να ελέγξουμε με επικοδομητικό τρόπο την πρόταση αυτή και ενδεχομένω να κάνουμε και προτάσει βελτίωση. Μία ερώτηση έχω να κάνω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση από πλευρά των Πρασίνων και από, τον, από τους επικριτές αναφέρθηκε ότι το πρόβλημα αυτό δεν θα επιληθεί με την πρόταση γιατί η υπερπληθώρα που έχουμε σήμερα ό,τι και να γίνει θα παραμείνει ενδυμική στο σύστημα και μετά το 2020 και αναφέρθηκε ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίσει με το στόχο αυτό το 40% μέχρι το 2030, το στόχος αυτός ουσιαστικά θα περιοριστεί στο 33%. Δεν εκεί θεωρώ αυτό. Μόνο και μόνο, δηλαδή, επειδή, επειδή η πολιτική του κλίματος δεν περιλαμβάνει μόνο το εμπόριο ρήπων, έχουμε και το effort sharing και Μόνο και μόνο γι' αυτό λοιπόν δεν στέκουν οι υπολογισμοί. Παρ' όλα αυτά να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ελέγξει αυτό το επιχείρημα και να μας πει κατά πόσον στέκει το γεγονός ότι τα πιστοποιητικά και μετά το 2020 θα παραμείνουν στην αγορά ή κατά πόσον ε, βελτιώνεται αυτό με την πρόταση την παρουσία αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος, και επόμενος είναι ο κύριος Μπάς Αχιάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την συγκεντρία κυρία Εικονή για την εισαγωγή, για τη συζήτηση, η οποία θα γίνεται ασφαλώς, θα συνεχίσει και μετά τις εκλογές για το αποθυματικό για τη σταθερότητα της αγοράς θα πρέπει να πω το εξή. Εμείς ως πράσινοι είμαστε κάπως απογοητευμένοι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μόνο αυτά που προτείνει. Γιατί έχουμε κάποια μεγάλα βασικά προβλήματα με το ETS ε και όλοι συζήτησαν το θέμα του backloading, το οποίο μας κερδίζει κάποιο χρόνο γιατί ο χρόνος στέδει διαρκώς. Για να γίνει πιο σωστή συζήτηση για μεταρρύθμιση του ETS, ε σωστή μεταρρύθμιση του ETS. Ε ως τώρα λοιπόν έχουμε δει μόνο αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ότι έχει πολλά ακόμα που προτείνει να ε, προτείνει για να επιλύσει το θέμα. Αν επικεντρωθούμε όμως το θέμα του αποθυματικού σταθεροποίηση τη αγορά, είναι ένα κλασικό παράδειγμα μια λύση, η οποία είναι υπερβολικά καθυστερημένη, κοίτοντας την μελέτη αντικτύπου της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση αυτή και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κοιτάει μόνο αυτό το πακέτο. Θα θέλαμε όμως να το κάνουμε. Αν υπάρχει λοιπόν ε, πλεόνασμα πιστοποιητικό 2 εκατομμυρίων τώρα και αυτό αυξάνεται και θα αυξηθεί μέχρι το 2,6 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020. Είναι τεράστιο το ποσό αυτό ακόμα και αν κοιτάξουμε και το σενάριο αναφοράς και πάλι συζητάμε για πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ε, τέτοιων αδειών. Και φυσικά θα μπορούσε να βοηθήσει το θέμα του αποθεματικού σταθεροποίηση, αλλά όχι και τόσο πια. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει κάτι παραπάνω για τη συζήτηση τώρα για το αποθεματικό αυτό. Φυσικά η συζήτηση θα εστιαστεί στο ποιου κανόνες ε, θέλουμε να δούμε για το πώς μπαίνουν όσοι άδειε μπαίνουν στο παθηματικό και τι θα γίνει μέχρι το 2021. Έχουμε τεράστιο πλεόνασμα τώρα. Γιατί λοιπόν να περιμένουμε και πάλι και να μην ξεκινήσουμε άμεσα με την επιβολή, επιβολή για τους κανόνες, για το πώς αυτό θα γίνει, πώ θα συμπεριληφθεί το μαθηματικό. 12% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε σε τίσιο επίπεδο. Περίεργο αυτό, γιατί 12%. 12,3% γιατί όχι. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σαφείς δεδομένου και του τεράστιου πλεονάσματος σε ό,τι αφορά το αποθυματικό σταθεροποίηση. Εγώ θα έλεγα τουλάχιστον 15%. Και αν απαλλάσσουμε τέτοια ποσά θα λέγαμε το ίδιο ποσοστό, 15% των αδειών που είναι σε κυκλοφορία να αφαιρεθούν. Και θα πρότεινα επίσης 300 ε, εκατομμύρια, όχι 400 εκατομμύρια είναι σημαντικοί αυτοί οι κανόνες, αλλά και πάλι, πρωτού ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για τους ακριβείς κανόνες, θα πρέπει να ξέρουμε τι επιπλέον μέτρα πρέπει να αναμένουμε, γιατί από δικής μας πλευράς είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και ένα μόνιμο πόσο το οποίο θα τύφεται στην άκρη. Τα πιστοποιητικά, οι άδειε που αφαιρούνται δεν θα πρέπει να επανειλησέρχονται σε καμία περίπτωση. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε το τι μπαίνει στο αποθεματικό σταθερότητα. Θέλουμε λοιπόν πιο πολύ σαφήνεια από την Ευρωπαϊκή, Επιτροπή. Ιδάλλως πώς θα αποφασίσουμε και για το αποθεματικό σταθεροποίησης. επιγόντως λοιπόν, σαφήνεια και ε, επιτέλους και λίγο παραπάνω φιλοδοξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, στι 12.30 πρέπει να προεδρεύσω μια συνεδρίαση, οπότε μάλλον δεν θα ακούσω την απάντηση. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω πάλι την ε, Σοφία Κονή για τι δικέ τη ε, παρατηρήσει. Οπότε λοιπόν ως ρυθμιστικός μηχανισμός για να λειτουργήσει το σύστημα ETC ε και να λυθούν κάποια προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν, κανείς δεν θα έχει αντίρρηση, είναι λογική η ρύθμιση. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με το σύστημα αυτό και όποτε αυτό έρχεται στο Ευρωκοινοβούλιο, ολόκληρο το ζήτημα του ETS ε ανακύπτει και φαντάζομαι και το στο μέλλον θα επανέλθει. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο προβλήματα που έχουμε και με το backloading θα έχουμε πάλι εδώ. Τώρα, ο στόχος αυτού του συστήματος είναι να εξασφαλίσει την μείωση των εκπομπών Ε, ε, της τάξης του 1,74% ετησίως. Ωραία. Όμως στο έγγραφο που εισάγει τον μηχανισμό, η Κομισιόν τονίζει ότι το, ότι το θέμα της τιμής είναι πολύ βασικό, γιατί είναι σημαντικό να δοθεί μια τιμή στον άνθρακα. Όσο το σκέφτομαι, όσο περισσότερο, τόσο περισσότερο πιστεύω πως εφόσον δεν δίνεις μια τιμή στον άνθρακα, δεν μπορείς να προχωρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και να ενθαρρύνεις ε, τις επενδύσεις σε επενδύσεις τις μάλλον σε χαμηλή εκπομπή άνθρακα. Όμως όταν μιλάμε για τιμή και τι επίπτωση θα έχει αυτό, τότε γίνεται ο χαμός, ε, γίνονται θάλασσα τα πράγματα και ο ένας αρχίζει να κατηγορεί τον άλλον. Έχει εκτιμηθεί και έχω δει διάφορους υπολογισμούς ότι αυτός ο μηχανισμός περίπου το 2020 θα αυξήσει τη τιμή των αδειών του άνθρακα κατά το ίμιση. Φαντάζεστε ότι πολλά λόμπι θα πούν ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά και η οικονομική κατάσταση ελπίζουμε ότι σε μια δεκαετία θα είναι βέβαια καλύτερη, αλλά θα αρχίζουν να κλαίγονται ότι δεν μπορούν να δεχτούν και να αντέξουν 30% αύξηση στην τιμή. Εφόσον λοιπόν θα γίνει αυτή η μάχη, γιατί να μην κάνουμε όντω τη μάχη, γιατί να μην το αναδιαρθρώσουμε τελείω το ETS και να αναγνωρίσουμε τα βασικά του μειονεκτήματα, αφού είναι το βασικό μέσο που έχουμε για τις ε, κλιματικές μας ε, πολιτικές. Γιατί το αφήνουμε μέχρι το 2020 και δεν το κάνουμε από το 2017, οπότε και θα μπορούσε να εισαχθεί αυτός ο μηχανισμός ε, γιατί τι... Μάλλον, τι γίνεται με τις προτάσεις για τη μεταφορά των ε, ε, αδειών backloading. Γιατί όχι, αφού έτσι και θα γίνει ο τσακωμός για τη μελλοντική κατεύθυνση της κλιματικής πολιτικής μας, ας αρχίσουμε από τώρα, ας ασχοληθούμε με την ουσία και ας ε, μην χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους κοσμητικούς, ε, τις κοσμητικές αλλαγές στο σύστημα που είναι χρήσιμες αλλά που δεν αντιμετωπίζουν το βασικό μας ζήτημα ότι δηλαδή πώς θα προωθήσουμε τις επενδύσεις σε ε, τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατάλαβα τις και άκουσα πολύ προσεκτικά τις εξηγήσεις της συναδέλφου Σοφία Κόνη. Άρα λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει για να εγγυηθεί την προβλεψιμότητα για την περίοδο 2021-2030 να δημιουργήσει αυτό το απόθεμα σταθερότητας της αγοράς που ε, θα λειτουργήσει σε ένας μηχανισμός με βάση στόχους και κανόνες επί τη βάση των οποίων οι όγκοι ε, θα προσαρμόζονται αυτόματα με υπόρους που θα προκαθορίσουμε. Δηλαδή δεν θα περνάμε πια από την νομοθετική διαδικασία για την προσθήκη και την αφαίρεση ποσοστώσεων και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτό το απόθεμα σταθερότητας λοιπόν της αγοράς θα είχε ως έργο το να θέσει σε λειτουργία μια προσαρμογή των όγκων των ποσοστώσεων όταν θα, αυτές θα βγαίνουν από μια συγκεκριμένη κλίδα. Εγώ ναι, συμφωνώ να προχωρήσουμε και όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Όμως, Ήδη ορίσαμε πιο φιλόδοξους στόχους περιορισμού των εκπομπών μέχρι το 2030 και θα πρέπει να θυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως δεν μπορεί να ξεχνά την πτυχή της ανταγωνιστικότητας στον ορισμό της ενεργειακής της πολιτικής. Οι προσπάθειες μείωση των εκπομπών που έγιναν το 2008 ήταν πολύ λιγότερο δαπανηρές από ότι αυτές που θα χρειαστεί να γίνουν από το 2020 και μετά μέχρι το 2030. Γιατί αυτά που ήταν αρκετά εύκολο να ξεκινήσουν ως πρόοδος έγιναν. Ενώ οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξή είναι πιο δύσκολες και πιο δαπανηρές σίγουρα. Οπότε ο μηχανισμός σταθερότητας όπως προτείνεται περισσότερο φαίνεται να έχει στόχο να βάλει σε απόθεμα τις ποσοστώσεις και όχι να σταθεροποιήσει τις τιμές και να θυμίσουμε ότι το ETS θα πρέπει να προσαρμόζεται στις κανόνες αγοράς και ότι δεν πρέπει να δυσκολέψει τη μεταπητική βιομηχανία ή όσους εξαρτώνται εντατικά από την ενέργεια. Αυτοί οι τομείς θα πρέπει να μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμη ορατότητα και να μην φέρουν οι ίδιοι το κόστος ε, της απανθρακοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. είναι το 11% των παγκοσμίων εκπομπών, οι εκπομπές μας και γι' αυτό μάλιστα χαίρομαι με την πρόσφατη απόφαση για σταθεροποίηση των κριτηρίων για την αναθεώρηση του καταλόγου των τομέων που εκτίθενται στις διαρροές άνθρακα. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο με βρίσκει σύμφωνη περισσότερο. Ήθελα λοιπόν να σας εκθέσω αυτές τις επιφυλάξεις και να πω προσοχή. Ας μην ακολουθήσουμε έναν δρόμο που θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολος για την οικονομία μας. Η κυρία Χίμπνερ. Ευχαριστώ. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών ε, είναι ένα στοιχείο της αγοράς που έπρεπε να λειτουργήσει καταπληκτικά. Το backloading ε, επίσης έπρεπε να αποκαταστήσει μια σταθερότητα των ε, τιμών. Ήταν σαν να βλέπαμε την αρχή του παραδείσου και τελικά ένα σύστημα που μεμονωμένα θα έπρεπε να φύγει από την αγορά ε, φεύγει τελείως, δημιουργούμε ένα τεχνητό σύστημα ε, προσπαθούμε να κινήσουμε κάποια νήματα αλλά τελικά ε, τι δίκαιο προβλέπουμε για, τα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τι δίκαιο είναι αυτό και τι νομοθεσία είναι αυτή που αλλάζει κάθε τρεις και λίγο. Και Πώς θα προβλέψουν αυτοί οι άνθρωποι τις, ε, τις επενδύσεις τους. Ούτε τις τιμές ε, δεν ξέρουμε και γιατί λέγαμε ότι ήταν τόσο καταπληκτικό το backloading αφού δεν ξέρουμε πώς να λειτουργεί. Υποτίθεται θέλαμε να σώσουμε το περιβάλλον, αλλά να δούμε με τι τρόπο θα το κάνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε την εντύπωση ότι τα έχουμε χάσει τελείως, τα έχουμε χαμένα, τα έχουμε παλαβώσει. Ναι. Κοιτάξτε, το ETS ε δεν είναι μια επίσημη αγορά και το να παρεμβούμε ε, σημαίνει ότι παρεμβαίνουμε στις ε, αγορές όπως παρεμβαίνουμε στις υπόλοιπες. Γιατί δεν μπορούμε να παρέμβουμε λοιπόν για το ETS αν δεν λειτουργεί. Η πρόταση, αυτή αξίζει να την εξετάσουμε και σε ό,τι αφορά και τις προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνούμε πάντα σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν και ελάχιστα όρια για τις τιμές. Αυτό θα μπορούσαμε να το α, αντιγράψουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, νομίζω ότι πρώτη, από 1η Απριλίου υπάρχει ε, μια σχετική πρόβλεψη στον Ε. Βασίλειο. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια καλή ιδέα και μπορούμε να σκεφτούμε κατά πόσο θα μπορούσε να εισαχθεί και μια μέγιστη τιμή προκειμένου να έχουν ένα μπούσουλα και όλες οι εταιρείε και να μπορούν να κάνουν το πρόγραμμά του. για να ξέρουν δηλαδή ελάχιστη και μέγιστη τιμή. Αυτό θα μπορούσαμε λοιπόν να το εισαγάγουμε σε ό,τι αφορά το backloading. Αυτό ήταν εξ αρχής σαφές ότι μόνο χρόνο θα μας κέρδιζε. Να δούμε τι θα κάνει και το επόμενο κοινοβούλιο, πώς ε, θα διαμορφωθεί η σύνθεση. Και τώρα λοιπόν θα ήθελα να ακούσω και την κυρία Σλίνγκερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνάδελφη Καρδίνη. Η συνάδελφος Γκαρδίνη, γιατί έχουμε φτάσει ήδη στις 12 η ώρα. Θα είμαι πολύ σύντομα, μη Πρόεδρε, γιατί οι συνάδελφοι ήδη ε, έχουν αναφέρει τα όσα σκέφτομαι και εγώ. Ανησυχώ πολύ για αυτή την Ευρώπη που συνεχίζει να υποβάλλει προτάσεις που θα επιβαρύνουν υπερβολικά Τη ε, νομοθεσίας. Αφού έχουμε μέχρι το 2020 αυτό το στόχο να αυξήσουμε το ΑΕΠ της μεταποιητικής βιομηχανίας που, έχει, ε, ε, που σήμερα βρίσκεται στο 14% και θέλουμε να το φτάσουμε στο 20%. Εγώ πιστεύω πως αυτός είναι ο χειρότερος τρόπος για να αρχίσουμε να επιδιώκουμε αυτό το στόχο που πρέπει να έχει την απόλυτη προτεραιότητα γιατί βλέπουμε μια ήπειρο που απεριμώνεται και κατά συνέπεια χώρες όπου η εισρωή των πολιτών για τις επόμενες εκλογές πέφτει στο 20% και μάλιστα αρχίζει να γίνεται αποδεκτό το 20%, το 30% πιθανή επιτυχία. Κάτω από το 20% καταστροφή. Εγώ πιστεύω πως αυτά τα ποσοστά συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στις ευρωεκλογέ θα είναι η οριστική καταδίκη της Ευρώπης που εξακολουθεί να μην αλλάζει πορεία. Μια Ευρώπη που πάει, κουτουλάει στον τοίχο και εξακολουθεί να σκέφτεται ότι είναι η πρώτη και καλύτερη ενώ είναι ε, η καταστροφή αυτή των οικονομιών και των χωρών που λειτουργούν ε, στη μεταπίση. Γιατί ναι, η Μεγάλη Βρετανία έχει το City και μιλάει για πράγματα που αν εμείς τα λέγαμε πριν από 20 χρόνια στους πολίτες μας θα είχαν σκάσει τα γέλια. Ε, και αν εγώ μιλήσω για οικονομία και για επιχειρήσεις και για μεταποίηση, μεταπητική βιομηχανία και αν μιλήσω για οροφές, για ελάχιστες τιμές, μιλώ στην ουσία για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν συνεννοούμαστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν να το ξανασκεφτείτε. Είμαστε στην αρχή. Ας σκεφτούμε εις βάθος και συνολικά. Γιατί δεν μπορούμε να Μιλάμε ο καθένας για το δικό του τομέα. Όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λέμε ότι είναι η δομή και ο ιστός της υπήρου μας και θέλουμε να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν. Αλλά αυτό το 20% του ΑΕΠ που, που παράγεται από τη μεταποίηση, αν ε, ε, με αυτή την περιβαλλοντική πολιτική το συνοδεύσουμε και ξέρω ότι είναι προτεραιότητα, δεν θα μπορέσουμε έτσι να επιτύχουμε αυτού του στόχου, που είναι θεμελιώδεις για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ευημερία και θέσει απασχόλησης για του πολίτε μα που εξακολουθούν να υποφέρουν από τι μετεκαταστάσει, από την απώλεια θέσεων εργασία και ανταγωνιστικότητα. περιβάλλον και βιομηχανία πρέπει να συνδυάζονται, αλλά αυτή εδώ η προσέγγιση είναι απόλυτα λάθο Ας το σκεφτούμε ε, ευρύτερα, πιο ανοιχτά. Σας ευχαριστώ κύριε Γκαρδίνη. Τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm. Αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς, ε, παρά το γεγονό ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και εσάς και την Επιτροπή Περιβάλλοντος και όλο το Κοινοβούλιο για την επιβράχυνση της περίοδου backloading, γιατί αυτό μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το backloading από την προηγούμενη εβδομάδα και να αποκτήσουμε και λίγη εμπειρία σε ό,τι αφορά το backloading. Το γεγονό ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή μα έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να συζητάμε τα δοσιατικά μέσα τα οποία έχουμε επιτάπητο τώρα και αυτά είχαν ζητηθεί και στη συζήτηση για το backloading και για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο του 2030 ασφαλώς συζητάμε και άλλα. Άλλες προσαρμογές στο ETS σε ό,τι αφορά τη μείωση του συντελεστή ε, γραμμικής σε ό,τι αφορά το 2030 και αυτή η αλλαγή επίσης θα βοηθούσε να ε, μειωθεί αυτή η αστάθεια που υπάρχει στο ETS. Δεν θα αρκούσε ωστόσο και η μελέτη αντικτύπου για το πλαίσιο 2030 και για το αποθεματικό καταδεικνύει με σαφήνεια αυτό το γεγονός. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ε, και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο στις συζητήσεις μας, γι' αυτό λοιπόν υπέβαλε αυτή τη νομική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θεματικό σταθεροποίηση της αγοράς ελπίζουμε να εγκριθεί γρήγορα στα τέλη του έτους. Έγιναν πολλές διαβουλεύσεις και τις προτάσεις αυτές με τους εμπλεκόμενους φορείς. Εξετάσαμε διάφορες δυνατότητες και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζήγησε όλους τους παράγοντες που προέκυψαν από τη διαβούλευση. Ένα από τα βασικά θέματα της πρότασης είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ρυθμιστική βεβαιότητα και σαφήνεια σε ό,τι αφορά το 2020 και το σχετικό πλαίσιο, προκειμένου όλοι οι φορείς του ETS να έχουν ένα διάστημα προσαρμογής προτού επιβληθούν αλλαγές για το παθηματικό σταθερότητα. Και γι' αυτό λοιπόν προτείναμε να εισαχθεί το 2021. Ωστόσο, όπως είπε η κυρία Οκόνη, με μια διάταξη που λαμβάνει υπόψη την ενδεχόμενη επανεμφάνιση των διατάξεων για το backloading στην τρίτη φάση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παραμείνουν τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο, σταθερότητα, πιο σταθερά για την τρίτη φάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση ότι θα υπάρχουν αυτές οι λίστες σταθερότητα, ε, νομική βεβαιότητα στη φάση 3. Γιατί τώρα δεν επισήλθαμε και δεν εξετάσαμε άλλες δυνατότητες που είχαν συζητηθεί με τους εμπλεκόμενους φορείς. Για παράδειγμα, μια τράπεζα άνθρακα. Στις συζητήσεις αυτές λοιπόν κατά στις σαφές είναι ότι το λιγότερο που ζητούν είναι μια διεκδικότητα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σαφές στις συζητήσεις για το backloading. Οι συζητήσεις ε, προκάλεσαν μεγάλη αστάθεια στην αγορά, ενώ η αγορά θέλει ουσιαστικά ένα όσο το δυνατόν πιο προβλέψιμο σύστημα γίνεται. Οποιαδήποτε τράπεζα άνθρακα θα είχε ε, έναν ε, εγγενή παράγοντα διακριτικότητας σε ό,τι αφορά και τις σχετικές συζητήσεις η τιμή η ελάχιστη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για έναν οικονομικό μηχανισμό, έναν μηχανισμό της αγοράς, όπως είπατε. Παρεμβαίνουμε στις αγορές, αλλά παράλληλα, αν θέλουμε να ορίζουμε όρια, και όρια και ανώτατα όρια στις τιμές, ουσιαστικά αφαιρούμε τον παράγοντα της ευελιξίας ε, από την αγορά και αυτό θα πρέπει να το δούμε και εν ώψη της κρίσης. Είναι φυσιολογικό ένα τέτοιο σύστημα να προσαρμόζεται στην οικονομική πραγματικότητα, στη μείωση της ε, ε, οικονομικής δραστηριότητας. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτό θεωρείται και ένα από τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Το γεγονός ότι υπάρχει ανταπόκριση των τιμών και διακύμαση των τιμών. Ιδάλλως ε, το κόστος ήταν πολύ πιο μεγάλο και για τους συμμετέχοντες της αγοράς και για τους παρόχους. Το γεγονός λοιπόν ότι έπεσε η τιμή είναι κάτι θετικό. Ετέθησαν ερωτήματα για μια πραγματική μεταρρύθμιση και πότε θα ήταν δυνατή αυτή. Είναι σαφές ότι καταρχάς θα πρέπει να κοιτάξουμε άλλα θέματα για το ETS μετά το 2020. Αυτό είναι τμήμα της συνολικής συζήτησης για τους ε, ορίζοντες και το πλαίσιο του 2030. Και πάλι σε ό,τι αφορά το 2030 δεν είναι μόνο το θέμα το ETS. Φυσικά ο στόχος για το 40% θα πρέπει να μεταφραστεί και σε στόχους που δεν καλύπτονται από το ETS και νομίζω ότι αυτό απαντάει τις ερωτήσεις του κυρίου Λίζε σε ό,τι αφορά το 40%, το 33%. Φυσικά θα έρθουν και οι άλλοι κλάδοι πέρα από το ETS και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 33% με τη συμπερίληψη άλλων μέτρων. Αυτό όμως είναι λίγο υποθετικό γιατί θα σήμαινε ότι θα αυξάνονταν τόσο πολύ οι εκπομπές που θα εξαντλούνταν το αποθεματικό. Εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ καλιστικό αυτό το επιχείρημα. Άλλες αλλαγές για το ETS. Όπως σας είπα, θα μπουν στο πλαίσιο των συζητήσεων για το 2030 και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με τη συγκεκριμένη πρόταση, που είναι μια σχεδιαζόμενη αλλαγή. Ένα μέτρο χωρίς ε, μεταμέλεια. Είναι ουδέτερο σε ό,τι αφορά το ΚΑΠ, δεν επηρεάζει το επίπεδο της φιλοδοξίας. Θα το συζητήσουμε αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας για το ETS ε και για άλλα στοιχεία στο πλαίσιο του 2030. Θα συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών και κυβερνήσεων αρχηγών κρατών κυβερνήσεων και θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένε νομοθετικέ προτάσει. Η πρότασή μα θεωρούμε ότι είναι μια πρόταση που θα ακολουθήσει την πορεία τη, δεν προκαλεί προβλήματα. Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα για μετά το 2020 και το μεταξύ εκτιμούμε ιδιαίτερα τα πέρα αυτή την πρώτη συζήτηση σήμερα για να συζητήσουμε τι λεπτομέρειε τη πρόταση για την σταθερότητα τη αγορά, τα όρια, του κανόνε, το πώ θα δημορφωθεί στην πράξη. Δεν θα επικεντρωθώ λοιπόν για το, στο γιατί επιλέξαμε το 12%, γιατί επιλέξαμε τα συγκεκριμένα τα όρια. Κάποια στιγμή στο μέλλον πολύ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρο, ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας για σήμερα. Και η συνάδελφος έχει και το τρένο που φεύγει. Σας εύχομαστε ό,τι καλύτερα. Ναι, το ξέρω. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δούλεψε τόσο σκληρά και θα δουλέψουμε πιο σκληρά και την επόμενη περίοδο. Ελπίζουμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα, τα λέμε στις 3. Στις 3. Και να ευχαριστήσω και τον Τζερμινή για την υπομονή του.